Cominciamo, cominciamo i nostri e Αρχίζουμε με τις ε, απογευματινές μας εργασίες. Έχουμε μαζί μας τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον καλωσορίζω. Ήταν και μέλος σε αυτή την Επιτροπή για πέντε χρόνια στην προηγούμενη θητεία και ξέρω ότι είχε ε, εργαστεί πολύ σκληρά. Θα μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της Ενέργειας που ε, ανέκυψε μετά από μία μελέτη. Είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική που θα μας βοηθήσει έτσι ώστε να προωθήσουμε μία ολοκληρωμένη πολιτική ενέργειας. Έχετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, ε, νιώθω σας στο σπίτι μου μαζί με εσάς, μέλη της Επιτροπής Ήτρε, ε, γιατί κατά την προηγούμενη εφητεία συμμετείχα στην Επιτροπή σας σχεδόν σε όλες τις συνεδριάσεις, κάτι το οποίο είναι αδύνατον πλέον. Αλλά σε 1,5 χρόνο ελπίζω να είμαι πίσω μαζί σας, διότι ήδη ε, έχω εκπληρώσει το 1,5 χρόνο της ε, αρχικής μου θητείας. Θέλω να σας παρουσιάσω κάτι που μου φαίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον για το μέλλον της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχήν στην Επιτροπή Ήτρε, δηλαδή τη δική μου Επιτροπή. Γιατί έγινε μια αρχική εκκίνηση του προγράμματος, της πολιτικής αυτής ιδέας, χωρίς επεξηγήσεις. Άρα πρόκειται για μια πολιτική όθηση προς τα εμπρός της ε, κοινότητάς μας ως προς την ενεργειακή της πολιτική, χωρίς να δοθούν λεπτομέρειες. Θα ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε μαζί τις λεπτομέρειες και τι σκέφτεστε ως προς το σχέδιο αυτό, το πρόγραμμα αυτό. Είναι θετικό για την κοινότητά μας ή ε, είσαστε σχετικά επιφυλακτικοί. Θα ήθελα να το συζητήσω μαζί σας καταρχήν. Όπως ξέρετε, έληξε η ΕΚΑΧ, δεν υφίσταται πλέον, αλλά Ίσως θα πρέπει να ανατρέξουμε σε κάτι ε, που να φέρει τη μορφή μιας ε, πολιτικής για την ενέργεια, όπως ίσχυε 60 χρόνια πριν με τον άνθρακα και το χάλιβα. Ήταν κάτι που ανέκυψε, προέκυψε από την φαντασία των προπατόρων. Να έχουμε μια κοινότητα του άνθρακα και του χάλιβα 60 χρόνια πριν. Κάπως έτσι ανέκυψε η ιδέα. Γιατί ήταν κάτι που δεν είχε συμβεί στο παρελθόν. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει η ενέργεια ολοκληρωτικά, δηλαδή το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, η έρευνα, η καινοτομία. Επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε την έρευνα και στον πυρηνικό τομέα. Υπάρχει και είναι ιδιαίτερα υποβοηθητική. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλει μεγάλες προσπάθειες. Ο Επίτροπος Έτιγκερ είπε ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση ε, έτσι ε, ώστε να προωθήσουμε το δεύτερο ενεργειακό πακέτο. So Η εφαρμογή των στόχων που προϋπάρχουν έτσι μας είπε ο Επίτροπος Έτιγκερ. Είχαμε μεγάλα προβλήματα με την αμοιβαία κατανόηση, τη σχήμα δηλαδή ακριβώς θα λάβει το τρίτο κοινοτικό πακέτο. Και η Επιτροπή θα προβάλλει ένα νέο σχέδιο απόδοση ενέργειας το 2020, υποδομές ενέργειας, πυρηνικά απόβλητα και η δεύτερη έκδοση, αυτή θα είναι η δεύτερη έκδοση της δράσης στον ε, τομέα της ενέργειας, μέσα από διάφορες οδηγίες. Θα θυμόσαστε τον κανονισμό για την προμήθεια φυσικού αερίου. Θα ψηφιστεί κατά την ε, Ολομέλεια, στην Ολομέλεια σε δύο μήνες και την ψηφίσατε και εσείς, εμείς δηλαδή η Επιτροπή μας ε, λίγους μήνες πριν. Αλλά έχουμε περιορισμένους πόρους ενέργειας, όπως γνωρίζετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως έχουμε και έναν ολοένα διονγκούμενο ανταγωνισμό από τρίτους, γιατί θα έχουμε μεγάλη έλλειψη ενεργειακών πόρων στο μέλλον. Άρα σήμερα θα πρέπει να κατέχουμε ηγετικό ρόλο ως Ευρωπαίοι, όχι ως κράτη. Γιατί τα κράτη δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε παγκόσμια κλίμακα. Αν λάβουμε υπόψη τη Βραζιλία, την Ινδία, την Κίνα, που είναι ε, αναπτυσσόμενες χώρες. Άρα οι κρατικές προκλήσεις ε, δεν είναι αρκετές. Πρέπει να υπερβούμε αυτό το πλαίσιο και αντιμετωπίζουμε προβλήματα για την αντιμετώπιση των ενεργειακών θεμάτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό. Ίσως οι πολίτες να μην καταλαβαίνουν ε, την πολιτική μας, αλλά καταλαβαίνουν όταν δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι, ενεργειακοί πόροι, όταν δηλαδή δεν τροφοδοτούνται με ενέργεια. Θα πρέπει να συνεχίσουμε με τη διαφοροποίηση πηγών ενέργειας, τις ανανεώσιμες, την πυρηνική ενέργεια που είναι πολύ σημαντική τα βιοκαύσιμα, αιωλική, ηλιακή ενέργεια, μείωση εκπομπών με την χρήση των ε, ορυκτών καυσίμων, από τη χρήση ορυκτών καυσίμων, χρειάζεται μεγάλη έρευνα. Και υπάρχει ένα ε, πολύ ε, χαμηλό κατόφλι για την έρευνα για την καινοτομία. Θα πρέπει να προωθήσουμε την κοινή έρευνα, την κοινή καινοτομία, την καινοτομία από κοινού, τις ε, νέες τεχνολογίες και ούτω καθεξής. Και βεβαίως ε, θα πρέπει μέσω αυτής της διασύνδεσης να προετοιμάσουμε τις νέες αγορές. Πώς μπορούμε να αρχίσουμε όντας ε, πραγματιστές. Υπάρχουν τρεις προτάσεις ενίσχυση συνεργασίας μέσα στα πλαίσια των δικτύων αυτών διασύνδεσης, κοινό ταμείο χρηματοδότησης νέων τεχνολογιών. Θα θυμόσαστε το, σχέδιο, το στρατηγικό σχέδιο νέων τεχνολογιών. Δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση καθώς και ομάδες παροχής και προμήθειας φυσικού αερίου. Τι εννοούμε όταν μιλάμε για κοινούς προμηθευτές. Θα πρέπει να μην έχουμε 27 επιμερισμένες διαπραγματεύσεις με όλους τους ε, παραγωγούς φυσικού αερίου. Μπορούμε να βασιστούμε στην υπάρχουσα, στην προϋπάρχουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δούμε και το θέμα της εξωτερικής προμήθειας. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σωστή κατανομή πετρελαίου και φυσικού αερίου μεταξύ κρατών μελών. Η εκμετάλλευση και η αποθήκευση, οι υποδομές γενικότερα. Ίσως θα αντιμετωπίσουμε και ορισμένες νομικές δυσκολίες. Δεν είναι και τόσο σοβαρές εάν φτάσουμε του, στους στόχους της ε, συνθήκης της Λισαβόνας που μιλάει για αλληλεγγύη στον ενεργειακό τομέα. Είναι μια νέα προσέγγιση η ενέργεια ως ειδική περίπτωση στη συνθήκη της Λισαβόνας. Επίσης, οποιαδήποτε λύση και εάν προωθήσουμε, η κοινότητα αυτή της ενέργειας θα πρέπει να προβάλλει ένα opt-in έτσι ώστε να προσχωρήσουν όλα τα κράτη όταν είναι έτοιμα. Να έχουμε μια σταδιακή προσχώρηση μικρών ομάδων κρατών μελών. Αυτό πάντα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Βεβαίως θα ήταν καλύτερα να αρχίσουμε από κοινού. Αλλά αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα προσχωρήσουμε σε μικρές ομάδες. Η λύση θα ήταν η προσχώρηση εννέα κρατών μελών αρχικά. Και υπάρχουν τρία βασικά πλεονεκτήματα κατά την άποψή μου. Οι οικονομίες κλίμακας, καταρχήν, γιατί μόλις επέστρεψα από την Κίνα, λίγες μέρες πριν και ξέρουμε τι σημαίνει οικονομία κλίμακας. Έχουμε εικόνα γι' αυτό. Και αυτό μπορούμε να κάνουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να προωθήσουμε η οικονομία κλίμακας αν είμαστε ενωμένοι σε ενεργειακά θέματα. Για 500 εκατομμύρια κατοίκων. Η μεγαλύτερη οικονομία σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαστε καλύτεροι και από τους Κινέζους εσωτερικά θα βοηθούσε τα κράτη-μέλη να επενδύσουν σε αυτές τις ε, ιδιαίτερα δαπανηρές υποδομές για να ολοκληρώσουμε την αγορά ενέργειας. Και θα υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις προμήθειας ενέργειας. Και αυτό μακροχρόνια σε μια αγορά μεγάλης κλίμακας. Επίσης θα πρέπει να δώσουμε τα σωστά κίνητρα. για να χρηματοδοτήσουμε και την έρευνα και την ανάπτυξη, έτσι ώστε η ευρωπαϊκή οικονομία να είναι ανταγωνιστική στη παγκόσμια. Μιλάμε για πράσινη τεχνολογία, για διατήρηση ενέργειας και για την πυρηνική ενέργεια. υπάρχει κοινό πρόγραμμα ερευνών. Και επίσης ε, μιλάμε για οικονομίες ε, ε, κλίμακας έτσι ώστε να είμαστε μία μεγάλη εμπορική κοινοπραξία για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε κοινέ αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου με άλλους διαπραγματευτές, μειώνοντας την τιμή της δηλαδή να είναι ανταγωνιστικές οι οικονομίες μας. Αυτό θα ήταν ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Επίσης, ως προς σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με την Κίνα, αν ε, το επιθυμείτε, θα ήθελα να επεκταθώ και σε αυτό το θέμα, έτσι ώστε να μας απασχολήσει και στη βασική μας συζήτηση για την ενεργειακή ευρωπαϊκή πολιτική. Έχει σημασία να δούμε πώς έχει αυτή η διασύνδεση και συνεργασία με την Κίνα και τη ΗΠΑ γιατί επισκέφτηκα και της ΗΠΑ και το συζητήσαμε αυτό το θέμα και στις ΗΠΑ. Πώς να αντιμετωπίσουμε το θέμα της κλιματικής αλλαγής, γιατί το 80% των προβλημάτων που άπτονται του κλίματος άπτονται και της ενέργειας. να δούμε πώς θα υπάρξει αυτή η διάδραση με τις άλλες μεγάλες δυνάμεις. Αν ε, μου επιτρέπετε θα σας πω λίγα λόγια και για αυτό το θέμα. Αλλά ως προς την... αυτό που έχει σημασία είναι πώς να δούμε την ε- Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Κοινότητα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Grazie al Ευχαριστούμε Πρόεδρε για αυτή τη συζήτηση που ανοίγει με τη δική μας Επιτροπή, την Επιτροπή Ήτρε. Τώρα έχουμε χρόνο για μια ανταλλαγή απόψεων. Υπάρχουν πολλοί εγγεγραμμένοι, λέει η Πρόεδρος. Θα ήθελα να, είναι, να είστε σύντομοι, συνάδελφοι. Ο συνάδελφος ε, Έντσου, ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον πρόεδρο Μπούζεκ για τη σημερινή επίσκεψη. Θα πρέπει να σας ομολογήσω ότι είναι η δεύτερη φορά που ακούω αυτή την ιδέα από εσάς. Την πρώτη φορά την είχα ακούσει στο Στρασβούργο από τον κύριο Ζακ Ντελόρ. Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει σειρά ερωτήσεων που ανακύπτουν ως προς το θέμα αυτό. θα είναι σε θέση τα κράτη-μέλη να κατανοήσουν ότι για λόγους αλληλεγγύης θα πρέπει να κινηθούν από κοινού, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση στον ενεργειακό τομέα από κοινού δηλαδή. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι και τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα που είναι ύψη τη σημασίας. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε το συμφέρον του πολίτη. Αυτό θα πρέπει να δεσπόζει. Πώς θα λυθεί το θέμα των μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων. Θα κατανοήσουν την αλληλεγγύη ή θα προβάλλουν μια δική τους αλληλεγγύη κατά των πολιτών. Εμείς ως ε, πολιτικοί θα πρέπει να προασπίσουμε τα συμφέροντα των πολιτών και του τελικού καταναλωτή. Μία άλλη ερώτηση που υποβάλλουμε συχνά είναι πώς θα προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες, τους καταναλωτές δηλαδή, σε περίπτωση μίας κοινής πολιτικής ενέργειας, όταν υπάρχει μία ενιαία τιμή ανεξάρτητα από το κόστος ζωής σε κάθε κράτος μέλος, διότι υπάρχει ένα κοινωνικό κόστος το οποίο θα πρέπει να επομισθούμε. Υπάρχουν ε, πολίτες που έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν είναι ενεργειακά ανεξάρτητη στο μέλλον. Πώς θα επιβάλλουμε τις ε, εναλλακτικές τεχνολογίες. Θα πρέπει να είμαστε ε, ρεαλιστές και να ξέρουμε ότι εφόσον εξαρτόμαστε από μαζικές εισαγωγές στον ενεργειακό τομέα, θα πρέπει να καταδείξουμε άλλη λεγγύη και να μην δεχτούμε την επικουρικότητα. Ευχαριστώ. Είναι πολλές οι παρεμβάσεις, θα πρέπει να τις ομαδοποιήσουμε, Πρόεδρε, αν συμφωνείτε, τις αναπέντε. Ακόμα και περισσότερες, λέει ο Πρόεδρος. Ε, μπατσίτης, πρίγω. Μπατσίτης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε ουδής αμφιβάλλει σήμερα ότι η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική θα πρέπει να συντονιστεί περισσότερο. Χρειαζόμαστε κοινούς κανόνες οι οποίοι να είναι δεσμευτικοί για κάθε χώρα μέλος. Δεν αρκούν τα ευχολόγια. Χρειαζόμαστε μια κοινή θέση όλων όταν διαπραγματευόμαστε με τους εταίρους μας. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας όταν προβαίνουμε σε αγορές ενέργειας, καθώς επίσης και στη χρήση των υπόλοιπων πόρων. Ωραίοι είναι οι φιλόδοξοι στόχοι μας και οι ευχές και οι επιθυμίες, αλλά σήμερα έχω ορισμένε αμφιβολίες σχετικά με το εάν στο πρώτο στάδιο προς μια ενεργειακή κοινότητα θα πρέπει να ανήκουν μοναχά εννέα χώρες μέλη και οι υπόλοιπες μπορούν να εντάσσονται σιγά σιγά και εφόσον θα είναι έτοιμες για την κίνηση αυτή. Πάλι βλέπω εδώ να μην υπάρχει επαρκής αλληλεγγύη και έχω αμφιβολίες εάν θα κατορθώσουμε να φτιάξουμε μια ενιαία ευρωπαϊκή κοινότητα εδώ και όχι μια Ευρώπη πάλι δύο ταχυτήτων όταν φτιάξουμε ας μια λέσχη πρώτα λίγων χωρών, οι οποίες όμως δεν θα έχουν, μάλλον οι υπόλοιπε δεν θα έχουν τις ίδιες δυνατότητες και επομένως δεν θα υπάρχει αλληλεγγύη. Και οι οικονομικά ασθενέστερες χώρες, για παράδειγμα μεταξύ αυτών και οι βαλτικές, θα πληγούν δεν θα έχουν δηλαδή διαρθρωτικές ή οικονομικές δυνατότητες να ενταχθούν στην πρώτη αυτή ενεργειακή κοινότητα. Γι' αυτό νομίζω ότι χρειαζόμαστε ξεκάθαρες απαντήσεις σχετικά με το ποια μορφή θα λάβει αυτή η ενεργειακή κοινότητα και ποιες χώρες θα ανήκουν σε αυτήν. Ρίμπικ. Ευχαριστώ και ιδιαιτέρως τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, κύριο Μπούσεκ, που νομίζω ότι διέγνωσε ορθά ότι αυτό που χρειάζεται είναι να αποκτήσει ανεξαρτησία η Ευρώπη στην ενεργειακή της πολιτική. Καθώς επίσης και να παίξει ρόλο προτύπου παγκοσμίω. συχνά όταν συζητούμε για την δημιουργία νέων συνθήκων, συζητούμε πρώτα τη χρηματοδότησή τους. Τα έσοδα από τις δημοπρατήσεις των δικαιωμάτων εκπομπής διοξιδίου του άνθρακος μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για την χρηματοδότηση μιας τέτοιας συνθήκης, διότι οι πρόσοδοι από τις δημοπρατήσεις αυτές κυρίως προέρχονται βέβαια από τον χώρο των ορυκτών καυσίμων και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να γίνει αποτελεσματικότερη η χρήση και κατανάλωση αυτών των ορυκτών καυσίμων. Επίσης, είναι σημαντικό οι διαδικασίες εγκρίσεων και για την ενέργεια αλλά και για τη δημιουργία δικτύων να τοποθετηθεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε υποτήρηση όλων των κανόνων βέβαια, να μπορούν με ταχύτητα να διεκπεραιώνονται σχετικές διαδικασίες. Το κυριότερο είναι, εφόσον εξακολουθεί να ισχύει η συνθήκη Ευρατόμ, χρειαζόμαστε ένα αντιστάθμισμα στη συνθήκη Ευρατόμ. Χρειαζόμαστε δηλαδή ένα δεύτερο πυλώνα που να διασφαλίζει ότι δεν θα προωθείται μοναχά η Ευρατόμ, δηλαδή μόνο η ατομική ενέργεια, αλλά και οι υπόλοιπε μορφές ενέργειας, ισοδύναμα ώστε από τη μια μεριά να υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδοτήσεως και αφετέρου βέβαια η συνθήκη Ευρατόμ να συμβάλλει και στην προώθηση και των άλλων ενεργειών αλλά και των ενεργειακών δικτύων. Γι' αυτό λοιπόν χαιρετίζω την ιδέα σας αυτή και νομίζω ότι πρέπει να συζητηθεί και περαιτέρω στην Επιτροπή μας. το λόγο. Merci beaucoup. Euh, merci, monsieur, monsieur le Président, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, γιατί ήρθατε εδώ μεταξύ μας για να μας μιλήσετε για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Υπάρχουν δύο μείζωνα ζητήματα που μας διαχωρίζουν. Καταρχήν, οι ενεργειακές πηγές και η ρύθμιση της αγοράς. Το κοινό πρόγραμμα, ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενέργειας δεν είναι ευσεβής πόθος γιατί θα πρέπει να υποστηρίξουμε να μιλήσουμε μάλλον για την αύξηση της ε, τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας. Πώς θα το δεχτούν οι αγορές, δηλαδή πώς θα δεχτούν οι επιχειρήσεις μια κοινή αγορά όταν αυξάνεται η τιμή της ενέργειας άρδιν και όταν οι τιμές ε, ε κυμαίνονται συνεχώς. Υπάρχει ένα θέμα ενεργειακής πρόσμιξης, θα μπορούσαμε να πούμε. Πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό στα κράτη-μέλη και μεταξύ αυτών σε εκείνα που, δημιουργούν την, που χρησιμοποιούν την υδροηλεκτρική ενέργεια ή την πυρηνική. Πώς να τους εξηγήσουμε ότι θα πληρώσουν πολύ ακριβά την ενέργεια τη στιγμή που χρησιμοποιούν φυσικό, ε, φυσικό αέριο ή άνθρακα. Τέλος, οι ιδιωτικέ επιχειρήσεις ενέργειας δεν θα δεχτούν μία μείωση των ε, αρμοδιοτήτων τους, του αποφασιστικού τους ρόλου. Τι θα κάνουμε με τις κοινοπραξίες. Βεβαίως ε, θα ήθελα να σας υποστηρίξω σε αυτό το πολύ σοβαρό σας ε, διάβημα παρά τις αμφιβολίες μου. Και, κυρία Welcome an initiative. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την εξαιρετική σας αυτή πρωτοβουλία σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα δέσμι μέτρων για τις κλιματικές αλλαγές. Δεν έχουμε βέβαια κοινή στρατηγική όλων των χωρών μελών για την ενέργεια. Θα περιληφθεί, αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση, η φυστάμενη νομοθεσία για την ενέργεια σε αυτήν την πρωτοβουλία ενεργειακής κοινότητας. Δεύτερο, μπορείτε να επεκταθείτε λίγο περισσότερο στο ποια είναι τα πλεονεκτήματα εάν συναπαρτήσουν την κοινότητα αυτή σε μια αρχική φάση μόνο ένα μέρος των χωρών μελών. Και τι θα πει όταν θα είναι έτοιμες οι χώρες μέλη θα μπορούν να ενταχθούν. Τι θα πει θα είναι έτοιμες διότι θα είναι πρόθυμες και συμμετέχουν ήδη στη στρατηγική για την ενέργεια και για το κλίμα. Δεύτερο, έχετε συζητήσει ήδη την νομική βάση της πρωτοβουλίας αυτής. Εν τέλει, δύο σχόλια, θετικά νομίζω, αφενός η χρηματοδότηση εάν θα βοηθήσει αυτό όλες οι χώρες μέλη να έχουν χρηματοδότηση για όλα τα σχέδια, για τις υποδομές που θα χρειαστεί να δημιουργηθούν. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό, εάν θα το συνδυάσετε αυτό και με την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Η ενέργεια και η ανταγωνιστικότητα βαδίζουν χέρι με χέρι. Ευχαριστώ. Η πρώτη, μου ερώτηση μάλλον είναι πώς θα, πώς θα περιληφθούν μάλλον οι υφιστάμενες στρατηγικές στην πρωτοβουλία σας αυτή. Διότι έχουμε ένα μεγάλο αριθμό οδηγιών, ανακοινώσεων, στόχων, μια ολόκληρη δέσμη μέτρων για την ενέργεια. Με τον συνάδελφο Ζαντό κλείνει αυτός ο πρώτος γύρος ερωτήσεων και θα απαντήσει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, είναι μεγάλη μας τιμή που βρίσκεστε εδώ μαζί μας. επειδή είναι κάτι το έκτακτο, θα ήθελα να ρωτήσω υπό ποια ιδιότητα είσαστε εδώ ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή ως ε, ε, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μεγάλης μας Ευρώπης. Ίσως θα ήταν ε, σκόπιμο να μας το διευκρινίσετε αυτό. Βεβαίως θα πρέπει να εξευρεθούν οι πόροι για την έρευνα γιατί οι πόροι είναι πενιχροί και για την έρευνα και για τις καινοτομίες επί του παρόντος. Ξέρετε ότι το δημόσιο χρήμα δεν περισσεύει. Εσείς λέτε ότι πρέπει να υποστηρίσουμε κάθε μορφή ενέργειας, ε, πετρέλαιο, ε, ε, φυσικό αέριο, πυρηνική, δηλαδή μιλάμε για ένα πολύ ευρύ φάσμα. Τη στιγμή όμως που έχουμε λίγα μέσα θα πρέπει να καταρτήσουμε ορισμένες προτεραιότητες. Με το θέμα, το θέμα ίτερ μάλλον θα μας απασχολήσει αργότερα. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η κοινοτική συνεισφορά η οποία τριπλασιάζεται από 2,7 σε 3,5 ως προς το κόστος παραγωγής. το ίτερ μας ζήτησε να έχει πάνω από 2 δις ε, ευρώ μετά το 2012-2013. Με το δικό σας πρόγραμμα πιστεύετε ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να επενδύουμε μαζικά σε αυτόν τον τύπο ενέργειας και να επαναπροσδιορίσουμε ή να ορίσουμε άλλες προτε... να ορίσουμε άλλες προτεραιότητες και να κινηθούμε προς τις ανανεώσιμες. Δίνω το λόγο στον Πρόεδρο για να απαντήσει στην πρώτη ομάδα ερωτήσεων. Και θα ήθελα ε, εκ νέου να σας ευχαριστήσω διότι μας μιλήσετε για αυτή τη μελέτη πρώτα-πρώτα στη δική μας Επιτροπή. Αυτό δείχνει μεγάλη ευαισθησία προς τις εργασίες της Επιτροπής μας. Uh, thank you, Madam Chair. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καθώς επίσης ευχαριστώ όλους και όλους τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις σας. Βέβαια δεν μπορώ να σας απαντήσω ευθύς αμέσως σε όλες αυτές τις ε, παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Όπως είπα και πριν, πρόκειται για μια απαρχή συζητήσεως και υπάρχει μια μεγάλη, νομίζω, ομοιότητα με το τι συνέβη στη δεκαετία του 80 του προηγούμενου αιώνα με την ενιαία αγορά όταν αρχίσαμε να συζητούμε στη δεκαετία του 80 ε, την ενιαία αγορά και στις αρχές της δεκαετίας του 90 και που άλλαξε ολόκληρη η ατμόσφαιρα σχετικά με την ενιαία αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάστηκαν όμως να περάσουν 3-4 χρόνια με τον πρόεδρο τότε Ζακ Ντελόρ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν νομίζω κάποιες ομοιότητες με εκείνη την φάση. Γίνανε πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Προτιμώ να απαντήσω σε ορισμένες από αυτές ξεχωριστά, για να σας δώσω πιο συγκεκριμένες απαντήσεις. Αλλά ας δούμε τις πιο σημαντικές τα οικονομικά θέματα και το ποιες είναι οι προσδοκίες των πολιτών μας, όπως ρώτησε ο κ. Έντσιου. Βέβαια, μιλώ για οικονομίες κλίμακος. Ε, αντιλαμβανόμαστε τι θα πει κλίμακα. Και σε μεγάλη κλίμακα μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα και να μειώσουμε το κόστος. Από την άποψη λοιπόν αυτή η απάντηση θα είναι νομίζω ότι μπορούμε να αναμένουμε καλά αποτελέσματα. Εάν σκεφτούμε τους καταναλωτές που αυτή τη στιγμή δεν έχουν, δεν χαίρουν πλήρου ασφαλείας, προμήθειας ενέργειας, τουλάχιστον σε ορισμένε χώρε μέλη. Για τον λόγο αυτό και μόνο είναι καλό να κατευθυνθούμε προς εκείνη την κατεύθυνση. Επίσης, η καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Ε, και αυτή απαντά στις ερωτήσεις σας, διότι έχουμε πολλά προβλήματα σχετικά με την εφαρμογή τη του δεύτερου και του τρίτου δηλαδή ενεργειακού πακέτου. Επίσης ολοκληρωμένα ευφυή e e δίκτυα, τα οποία επίσης μπορούν να μας βοηθήσουν σχετικά με τις τιμές. Η κυρία Γκροστέτ ε, έθεσε ερώτηση σχετικά με τι τιμές. Δεν σημαίνει ότι οι τιμές θα είναι ίδιες. Είναι όπως και τώρα, ε, όπου κυκλοφορούν πολλά αγαθά στην ενιαία αγορά, δεν είναι όμως παντού με τις ίδιες τιμές. Θα είναι όμως δυνατό να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα που εντοπίζονται στον τομέα της ενέργειας μαζί. Για μένα το κρίσιμο θέμα είναι να δοθούν κοινοί πόροι για την τεχνολογία. Γιατί και οι τιμές εξαρτώνται από την τεχνολογία. Αν λοιπόν μπορούμε να αναπτύξουμε πολύ ευρύτερα και να χρησιμοποιήσουμε την πυρηνική ενέργεια σε ορισμένες χώρες τουλάχιστον μέσα σε συνεργασία, αυτό θα μας βγει φθηνότερο εν τέλει. Αλλού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αιωλική ή την ηλιακή ενέργεια. Ανταλλαγή όμως όλων των επιτευγμάτων και στον τομέα της τεχνολογίας και να δαπανούμε χρήματα μαζί για την ανάπτυξη τεχνολογίας και για την καινοτομία. Είναι το επόμενο βήμα μετά από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας ή το πρόγραμμά μας για την ανάπτυξη που θα αρχίσει να εφαρμόζεται σε λίγα χρόνια και αν προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο νομίζω είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να δαπανίσουμε τους πόρους πολύ πιο αποτελεσματικά. για τις ερωτήσεις του κυρίου Μπαλτσίτης. Κοινή διαπραγματευτική θέση. Λέτε ότι αμφιβάλλεται αν νέας, εννέα χώρες μέλη... Βέβαια δεν θα είναι καλή λύση ούτε για μένα. Είπα μόνο ότι οι εννέα χώρες μέλη θα πρέπει να είναι το ελάχιστο. Η συμφωνία των χώρων, εννέα χωρών μελών θα πρέπει να είναι το μίνιμουμ. Αλλά βέβαια και για μένα δεν είναι καλή λύση αυτή θα πρέπει να πράξουμε πάντο δυνατό ώστε να συμμετάσχουν όλες οι χώρες. Θα απαντήσω τι σημαίνει από την σκοπιά των νομικών επιλογών. Νομίζω ότι υπάρχουν τέσσερις. Μπορούμε να τροποποιήσουμε την συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ούτε καν μπορείτε να φανταστείτε πόσο δύσκολο θα είναι. Άρα μάλλον να εγκαταλείψουμε τη λύση αυτή. Δεύτερη λύση, ενισχυμένη συνεργασία. Είναι ο καλύτερος τρόπος στην βάση της συνθήκης της Λισαβόνας. Θα ήταν λοιπόν εάν όλες οι χώρες μέλη συμφωνήσουν σε μια ενισχυμένη συνεργασία και να φτιάξουν κάτι σαν μια ευρωπαϊκή ενεργειακή κοινότητα με ισχυρή πολιτική υποστήριξη. Και κατελάχιστον όρο 9 χώρε μέλη, που δεν θα είναι η καλύτερη λύση, καλύτερα 27 χώρε μέλη, να προχωρήσουν σε ενισχυμένη συνεργασία. Μπορούμε να εγκρίνουμε, νομομαθεί τα είπαν αυτά, πάντα στη βάση της συνθήκης Λισαβόνα, αλλά είναι η πιο προωθημένη λύση, μια συνεργασία για την ενέργεια. Και είναι απαραίτητο βέβαια να το συζητήσουν πρώτα οι νομομαθείς. Αν είναι δυνατόν να γίνει αυτό στην βάση της υφιστάμενης συνθήκης της Και επίσης μπορούν, μπορούμε να βασιστούμε σε ad hoc ρυθμίσεις, όχι βέβαια μακροπρόθεσμα αλλά βραχυπρόθεσμα με πιο μετριοπαθείς στόχους για ορισμένους, ορισμένους τομείς πολιτικής. Ε, εξαρτάται από ποιους τομείς πολιτικής θα θέλουμε να επιλέξουμε. Και αυτή λοιπόν μπορεί να είναι μια λύση να επιλέξουμε ορισμένους τομείς, όχι όλους. Ξαναλέω ότι πρόκειται για την αφετηρία μια συζητήσεως. Θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις σας και γραπτός και θα σας στείλω και τις σχετικές πληροφορίες, γιατί αρχίζουμε τώρα μια σοβαρή συζήτηση. Για τον κύριο Ρούμπικ τώρα. Η χρήση και παραγωγή ορυκτών καυσίμων και χρήση με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ασφαλώς είναι πολύ σημαντική. Ιδίως στην χώρα σας. Δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα εκεί. Γιατί δεν έχετε και πολλά ορυκτά καύσιμα. Αλλά γενικά το πρόβλημα είναι μέγα. Και πολλέ χώρε ανησυχούν για την υπερβολική χρήση των ορυκτών καυσίμων λόγω των θεμάτων του κλίματο. Και λαμβάνοντας υπόψη, όπω είπατε, όλε τι πιθανέ επιλογέ. Και βέβαια η Ευρατόμ που είναι καλό παράδειγμα της συνεργασίας και κυρίως στον τομέα της έρευνας. Τώρα πάλι ερώτηση κυρίας Γκροστέτ. Η πόροι είναι ένα πρόβλημα και η ρύθμιση της αγοράς είναι το άλλο πρόβλημα. Σωστό. Η ρύθμιση της αγοράς. Προσπαθήσαμε να κάνουμε στο δεύτερο και στο τρίτο πακέτο ενέργειας. Θα χρειαστούμε κάποια πολιτική όθηση, κάποια πολιτική υποστήριξη. Εάν βεβαίω αποφασίσουν όλες οι χώρες μέλη με τη συνεργασία του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν ότι θα θέλαν να προχωρήσουν σε ρύθμιση της αγοράς, μιας κοινή αγοράς, για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην ενέργεια, ας πούμε. Ίσως, ας πούμε, και για μείωση των τιμών. Όπως είπα πριν, που θα προκύψει από τις οικονομίες κλίμακος. Πώς ρωτήσατε να εξηγήσουμε στις χώρες μέλη, σε όλες τις χώρες μέλη, ότι αξίζει τον κόπο να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Έχουμε τρεις δυνατότητες. Ενίσχυση, ενίσχυση της συνεργασίας στα ενεργειακά δίκτυα, διότι καλύτερα ενεργειακά δίκτυα, ασφαλώς, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, κοινή πόρη για την έρευνα. Και αυτό ενδιαφέρει όλες τις χώρες μέλη, νομίζω. και της ανάπτυξης που είναι βασισμένη στο αέριο ή στο πετρέλαιο. Το πιο δύσκολο θέμα αυτό για όλους μας. Εάν είμαστε διατεθειμένοι δηλαδή να το πράξουμε, διότι τώρα μιλούμε και επιχειρηματολογούμε ξεχωριστά από το θέμα αυτό. ενώ θα έπρεπε να πάμε να συζητήσουμε με τους γειτονές μας, με τους προμηθευτές μας. Πάλι εννοώ με μία φωνή ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα ήταν μεγάλη πρόοδος αν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Βέβαια δεν είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσει να γίνει. Πάντως θα ήταν ε, σημαντικό για όλους μας. Και η κυρία Καλουάριο. Η υφιστάμενη στρατηγική και όσα αναπτύσσουμε τώρα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Κοινότητα. Αυτό για μένα δεν είναι πρόβλημα, διότι προσπαθούμε να αναπτύξουμε την ενιαία μας αγορά. Και πάλι μιλήσατε για την εμπλοκή ορισμένων χωρών μελών. Βέβαια, εγώ προτιμώ να είναι όλες για την νομική ε, βάση. Είπα, ε, ανέφερα τις τέσσερις δυνατότητες. Η πρώτη αποκλείεται βέβαια, ενώ την τροποποίηση, η αναθεώρηση της ε, συνθήκης Λισαβόνας, κάτι που είναι αδύνατον αλλά ίσως οι άλλες τρεις επιλογές είναι δυνατόν να εφαρμοστούν. Χρηματοδότηση βέβαια και χρηματοδότηση της υποδομής και της έρευνας. Είναι σημαντικά αυτά. Και μπορεί να γίνει πολύ ευκολότερα από κοινού. Η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας ενέργειας μιλούμε για ανταγωνιστικότητα στο παγκόσμιο επίπεδο, όχι μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι πολύ σημαντικό για μας λοιπόν να υπάρξει συνεργασία στην Ευρώπη, ώστε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί παγκοσμίω. Και η τελευταία ερώτηση σχετικά με τις προτεραιότητες. Αυτό είναι θέμα επιλογών. Δεν έχει κρυθεί. Εγώ έθιξα κάποιες προτάσεις, ανέπτυξα κάποιες προτάσεις. Ορισμένες είναι πιο εύκολες ή πιο βολικές για όλες τις χώρες μέλη, όπως για παράδειγμα εξοικονόμηση της ενέργειας, η καλύτερη αποδοτικότητα της ενέργειας, οι ανανεώσιμες ενέργειες, διότι γνωρίζουμε ότι αυτά είναι κρίσιμα για όλες τις χώρες η μέλη. Μπορούμε να πούμε επίσης ότι ορισμένες νέες τεχνολογίες όπως η αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακος, το φλέξι πρόγραμμα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, με υποδομές που ε, εν μέρει θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε αρχίσει λοιπόν σε ορισμένου τομεί τη συνεργασία και βαθιά συνεργασία. Δεν είναι βεβαίω δυνατά όλα. Μια όμως ισχυρή πολιτική όθηση με σημαντική πολιτική υποστήριξη υπέρ των διαφόρων κοινών δράσεων στον τομέα της ενέργειας, θα είναι το μέγα πλεονέκτημα, κατά τη γνώμη μου, της ευρωπαϊκής αυτής ενεργειακής κοινότητας και ίσως να ε, καταστήσει ευκολότερες τις λύσεις και για τις ευρωπαϊκές αγορές και για τους ευρωπαίους πολίτες. Διότι εν τέλει ε, υπέρ αυτών θα αποβεί, υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών, με καλύτερες τιμές, και μεγαλύτερη ασφάλεια προμήθειας. Και βέβαια και την προστασία του περιβάλλοντος. Τα τρία λοιπόν αυτά στοιχεία. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά υπόσχονται ένα καλύτερο μέλλον. Αυτά νομίζω για την ώρα. Πάντως λέω και πάλι Θα σκεφτώ πολύ σοβαρά όλες τις ερωτήσεις σας και θα απαντήσω και γραπτός σε ορισμένες, εάν, εάν θεωρήσετε ότι κάτι δεν απάντησα τώρα. Γιατί όπως είπα πρόκειται για την αρχή μιας ανοιχτής συζήτησης. Ας προχωρήσουμε στις επόμενες. Εννέα ομιλητές ζητούν το λόγο. Θα ήθελα να είσαστε ιδιαίτερα σύντομοι. Κλοντ Τούρμες. Ε, President Πρόεδρε Μπουζέκ, ομολογώ με κάθε σεβασμό ότι αυτά είναι πολύ ακατανόητα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω ακριβώ υπό ποια ιδιότητα μιλάτε εδώ. Δική σα ιδέα είναι γιατί ε, είστε μέλος τη ε, δικής μας Ευρώπης ή πώς, γιατί, για πέστε μας σε ποιο πλαίσιο εντάσσεται η παρέμβασή σας. Δεύτερον, έχοντα εργαστεί για νομοθεσία για την εσωτερική αγορά, για την ε, νομοθεσία για την αποτελεσματικότητα, για τι ε, ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, για την νομοθεσία για το φυσικό αέριο, ομολογώ ότι έχουμε αρκετή νομοθεσία, αρκετέ δυνατότητε. Αν θέλετε να κινηθείτε προ την αποτελεσματικότητα, καλώ γίνεται. Έχουμε 10, 12 ε, νομοθετικά κείμενα για να προχωρήσουμε. Το ίδιο και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για την εσωτερική αγορά, μόλις τελειοποιήσαμε κάποιες δέσμες μέτρων, αυτή τη στιγμή τελειοποιούμε επίσης την ε, οδηγία για την ε, ασφάλεια τροφοδότησης με φυσικό αέριο. Το να ξεκινά δηλαδή τώρα μία καινούργια μεγάλη ιδέα, πρέπει να ξέρουμε ποια θα είναι η αλληλένδεση μεταξύ αυτών των μεγάλων ιδεών στη συνθήκη με την πραγματική νομοθεσία που έχουμε στα χέρια μας ήδη. Όσοι δεν έχουν διαβάσει τις συνεχικές ε, εκθέσεις που βασίζονται, γιατί ε, που και που κύριε Βουζέκ εξεπλάγει, αλλά κάνετε δηλώσεις που ε, δεν αντικαταπίζουν καθόλου σε αυτή την έκθεση εδώ που είναι υποτίθεται η βάση όλων. Ας είμαστε λοιπόν ακριβείς και ας οργανωθούμε πιο στρατηγικά. Γιατί αλλιώς θα βλάψουμε αυτό που θέλουμε. Ε, ähm, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέει κυρία Νίμπλε, δύο παρατηρήσεις πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Καλό μου φαίνεται που ήρθετε εδώ για να πτύξετε κάποιες ιδέες. Είναι νομίζω κάτι που αρμόζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να τυπώνει κάποιες ιδέες. Και ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μας για να παρουσιάσετε τις δικές σας ιδέες, να τις συζητήσετε μαζί μας. Είμαστε ανοιχτοί για ιδέες, για προτάσεις και γι' αυτό μου φαίνεται ότι είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Έχω ορισμένε ερωτήσει. Ε, η μία αυτή στρέφεται προ εμά, ε, έχει υποβληθεί και γραπτά. Με εξέπληξε η ιδέα ότι εδώ πρόκειται για τη δημιουργία αμαθοποιημένων ε, αγορών για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Πώς το φαντάζεσαι αυτό δηλαδή. Εγώ έχω την εντύπωση ότι η ίδια η βιομηχανία οργανώνεται μόνη τη και πέρα από τα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν υπάρχουν ορισμένα οικονομικά πλεονεκτήματα, αν δημιουργηθεί κάποια ένωση για την αγορά των πηγών αυτών ενέργεια, νομίζω ότι οι ενδιαφερόμενοι θα το κάνουν. Ε, αναρωτιέμαι, τι θα κάνει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά, ποιο θα είναι πολιτικά το πλαίσιο που θα πρέπει να δημιουργήσουμε. Ίσως θα να συμπεριλάβετε και αυτή την ερώτηση. Ευχαριστώ, Οντί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ χαίρομαι που είστε εδώ. Καμιά φορά ε, σας βλέπω ε, δυσαρεστημένο στην Ολομέλεια. Εδώ σας βλέπω όμως πολύ ευτυχή και χαίρομαι. Θα ήθελα να πω στι γενικέ γραμμέ συμφωνώ με του στόχου σα. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα όμω στη λέξη κοινότητα. Αναφερθήκατε στην άνθρακα και χάλιβα. Αντί να κάνουμε δηλαδή να παράγουμε όπλα, παράγουμε οικονομία. Αυτή ήταν η μια Μετά είχαμε μια οικονομική κοινότητα, ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα και χρειάστηκε πολλού χρόνου για να περάσουμε στην Ένωση. Και σήμερα έχουμε μια, ένα νομικό πρόσωπο που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα να δημιουργήσουμε πάλι μια κοινότητα δεν ξέρω πως είναι προβληματικό. Και νομίζω ότι θα χαθούν τελείως οι, οι πολίτες και ορισμένοι βουλευτές ανάμεσα στα επίπεδα δράσης της κοινότητας, το διακυβερνητικό, την ε, τράπεζα στην οποία είναι μέλη τα κρατημέρια και ε, δεν ξέρουμε ποιος ηγείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος ελέγχει τι τα δάνεια στην Ελλάδα, δεν ξέρω τι είναι το κοινοτικό τμήμα, ποιο είναι το μη κοινοτικό τμήμα και μια που η συνθήκη της Λισαβόνης επιτρέπει σε κράτη-μέλη να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα γίνει αν φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση το κράτος αυτό και παραμείνει στη δική σας κοινότητα. Ποια είναι η πολιτική ομάδα στήριξη που έχετε για αυτή την πρωτοβουλία που είναι πάρα πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα. Οι ηγοί κρατών και κυβερνήσεων σας ακολουθούν. Ευχαριστώ. Η κυρία Πουδηματά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σε συνέχεια και του ερωτήματος του αγαπητού συναδέλφου του κυρίου Ντή, θέλω να πάω σε μια περισσότερο ε, αισιόδοξη εκδοχή κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι αν υπάρχει ένα βασικό συμπέρασμα από τις ε, συνθήκες κρίσης τις οποίες διάγουμε σήμερα είναι ότι ε, χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη και όχι λιγότερη Ευρώπη και με αυτή την έννοια χρειάζεται να συντασσόμαστε όλοι ε, πίσω από σχέδια που να μας ενώνουν περισσότερο και όχι να μας χωρίζουν. Άρα λοιπόν σε ό,τι αφορά αυτή την εξαιρετική κατά τη γνώμη μου πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ενεργειακής κοινότητας ε, θεωρώ ότι έχουμε κάθε λόγο και κάθε συμφέρον ε, να ε, υποστηρίξουμε τη σύνταξη του συνόλου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πίσω από την πρωτοβουλία αυτή και να προσπαθήσουμε να δεσμευτούμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να αποφύγουμε να δημιουργηθούν νέε διαχωριστικές γραμμές με κάποια κράτη-μέλη που θα προχωρήσουν και κάποια άλλα που θα έπονται. Ε, για να υλοποιηθεί όμω αυτό το εξαιρετικά φιλόδοξο ε, σχέδιο ε, υπάρχει μια εκ των όνου προϋπόθεση που αφορά στη δημιουργία σύγχρονων, αναβαθμισμένων διασυνδεδεμένων και αποδοτικών ε, ενεργειακών ε, δικτύων και ιδιαίτερα δικτύων που να υπηρετούν τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020. Ε, είπαν διάφοροι συνάδελφοι, υπάρχουν πολιτικές, επιμέρους, νομοθεσίες, προτάσεις, προγράμματα. Όλα αυτά είναι λίγο αποσπασματικά και μεμονωμένα και λείπει μια συνεκτική στρατηγική στήριξη στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τα δίκτυα, Θεωρώ ότι υπάρχουν τρει ισότιμοι πυλώνε που θα πρέπει να προωθηθούν και αυτοί αφορούν στην πρόθεση των ενεργειακών διασυνδέσεων, στην ε, αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό εφιστάμενων δικτύων, ιδιαίτερα στα νέα κράτη-μέλη, και βεβαίω στην πρωτοβουλία για την ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων που υποστηρίζονται ε, και στο πλαίσιο της στρατηγικής 2020. Ε, το ερώτημά μου, κύριε Πρόεδρε, είναι είναι δυνατόν όλα αυτά να υποστηριχθούν χωρίς δραστική αύξηση ε, των ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονται ε, για τη χρηματοδότηση των ε, ενεργειακών σχεδίων και το δεύτερο, μπορεί αυτή η αναγκαία ενιαία συνεκτική στρατηγική που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να υλοποιηθεί χωρίς ένα κοινό ευρωπαϊκό ταμείο που να συντονίζει όλες αυτές τις χρηματοδοτικές δράσεις για την πρόωθηση αυτού του σχεδίου. Ευχαριστώ. Ε, ε, ε, Πρόεδρε και κύριε Μπούζακ, αρχίστε την παρουσία σας τονίζω στην ανάγκη να ενδυναμωθεί η ισχύουσα νομοθεσία, παραδείγματο χάρη όσον αφορά τι οδηγίε για την εσωτερική αγορά. Θεωρώ όμω ότι αυτό το είδαμε σε πολλού άλλου τομεί. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε για να φτάσουμε μια πραγματική πολιτική, κοινή πολιτική ενέργειας. Εδώ συζητήσαμε για την οδηγία για τις πηγές και είχαμε το θέμα του κλίματος το 2015 και είπαμε τώρα θα είμαστε οι ηγέτες του κόσμου. Στην πραγματικότητα όμως τα κράτη-μέλη του COP15 έκαναν ο καθένας ό,τι ήθελε. Και ο ηγέτης ήταν ο Στάνισλα Λουμούμπα. Γιατί δεν ήταν ενωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την περασμένη εβδομάδα πήγα στο Καζαξάν σαν μέλο τη Αντιπροσωπεία Κεντρική Ασία και το Καζαξάν έχει επίση σχέσει με μονομένα μελη που προωθούν τα δικά του συμφέροντα. Θα ήθελα να ξέρω, γιατί αυτά γίνονται και στη Ρωσία, να ξέρω πώ βλέπουμε τη δυνατότητα να πειθούν τα κράτη-μέλη να έχουν ένα κοινό πλαίσιο για την αντιμετώπιση εξωτερικών της Ένωσης πηγών ενέργεια από τη Ρωσία ή από άλλες χώρες. γιατί ορισμένα κράτη-μέλη έχουν δικέ του καλές ε, συμφωνίες. Αλλά απέχουμε πολύ από μια κοινή πολιτική. Εσείς είπατε εισαγωγικά ότι θέλετε να υπάρχει κάποια κοινή αντίδραση και προς την Κίνα, γιατί είμαστε ανταγωνιστές της Κίνας, είδα στην Ινδία. Δια που ε, τι έγινε με το ουράνιο που το έλεγχαν οι Γάλλοι και τώρα η Κίνα προσπαθεί να μπει εκείνη στο παιχνίδι και να διώξει τους Γάλλους. Επίσης θα ήθελα να ξέρω ποιες είναι οι νέα χώρες μέλη που άρχισαν να συνεργάζονται μεταξύ τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τσίτσεστερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, Ιωζή, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μεγάλη χαρά να σας βλέπουμε πάλι σε αυτή την επιτροπή, τη δική σας επιτροπή στην τελευταία θητεία. Και θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου που διατηρείται επίσης στις συνδέσεις που έχετε με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ενέργειας, σαν πρώτος αντιπρόεδρος. Ζητώ συγγνώμη δεν ήμουν παρόν την όλη που κάνετε τη δική σας παρουσίαση, αλλά είχατε την καλοσύνη στην περισμένη σύνοδο του Στρασβουργού να έχετε κάποιο χρόνο διαθέσει να συζήσετε το θέμα με μένα. Χρειαζόμαστε όλοι να κατανοήσουμε σαφέστατα το τι υποβάλλεται αυτή τη στιγμή. Έχω την εντύπωση ότι δεν καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Αναρωτιέμαι ιδίω τι είναι το καινούριο. Προβλέπετε πλήρη αναθεώρηση και ονομασία και παρουσίαση της ευρωπαϊκής πολιτικής ενέργειας. Γιατί ήδη έχουμε πάρα πολύ ε, ενεργή πολιτική ήδη, όπως είπε και ο συνάλφος Κλωτ Τούρμες. Και παραδέχομαι ότι έχω κάποιες ανησυχίες όσον αφορά η πρόταση για τροποποίηση συνθήκης ή και νέες συνθήκες, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κουραστεί από συνθήκες πια. Και δεν ήταν καλό, νομίζω, να προσπαθήσουμε να ξαναξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία τόσο γλίγορα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τι ξεκινήσαμε στην ε, περασμένη θητεία ήδη. Και είναι να προχωρήσουμε προς την διάγουσα. Θα σας στηρίζαμε εκεί. Θα πρέπει επίσης να παραδεχτώ μία ανησυχία ακούγοντας μια ε, φωνή από το παρελθόν, ε, μια αναφορά στον ε, κύριο Ντελόρ. Ίσως είναι μια βρετανική ανησυχία αυτή, αλλά είναι μια ανησυχία. Ομολογώ ότι υπάρχει ένας κίνδυνος με την υποβολή νέων ε, πρωτοβουλειών ή νέων σφαιρικών πρωτοβουλειών ότι δηλαδή σταματάμε αυτό που κάνουμε και διακυβεύουμε τα πάντα και μεταξύ συζητάμε αυτές τις νέες ε, ε, πρωτοβουλίες και την ισχύουσα νομοθεσία. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε την συνθήκη της Λισαβόνας, όπου ο κύριο Κοκ, συγκεκριμένος Ολλανδός ε, πολιτικός είχε έρθει εδώ και είχε πει ότι 204 ε, πρωτοβουλίες είναι 200 παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Και δεν προχωρήσαμε. Το μόνο που πετύχαμε ήταν να προχωρήσουμε για την απελευθέρωση της ενέργειας, κάτι πάνω στο οποίο είχαμε ήδη από πριν αρχίσει να εργαζόμαστε. Από τότε που πήγα στο κοινοβούλιο εδώ, πριν από 16 χρόνια δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι προσπαθώ να πετύχω μια εσωτερική αγορά, μια ενιαία αγορά, απόλυτα απελευθερωμένη στον τομέα της ενέργειας. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί και πολλά θα πρέπει ακόμα να γίνουν σίγουρα. Αλλά Μόλις ξεκινήσαμε την νομοθεσία για την τρίτη δέσμη, θα πρέπει να δώσουμε αρκετό χρόνο για να μπορέσει να μεταφερθεί στην νομοθεσία των κρατών μελών, να εφαρμοστεί και να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Γι' αυτό χρειαζόνται χρόνια. Και αν δεν το κάνουμε αυτό, υπάρχει ο κίνδυνος να σταματήσει η τρέχουσα εργασία χωρίς να πετύχουμε τίποτα. Τελειώντας, θα ήθελα να προεδοποιήσω για κάτι, αν μου επιτρέπετε. Στο πρώτο δεύτερο κοινοβούλιο, ο τότε, η τότε Επίτροπος όλο το Παλάθιο, μας υπέβαλε μία πρόταση για τη διαχείριση των αποθεμάτων πετρελαίου. Μια εποχή που ανησυχούσαμε για την τροφοδότηση της παγκόσμιας οικονομίας με πετρέλαιο και η πρόταση ήταν να αλλάξει το καθεστώς για τη διαχείριση των αποθεμάτων που βασίζεται του IEA και να αλλάξει ο ρυθμός των ημερών από 90 σε 120 ημέρες από θέματα και να δώσει την ισχύ στην Κομισιόν να παρεμβαίνει στην αγορά για να εξομαλύνει τα πράγματα. Δηλαδή να πουλήσει από θέματα να αγοράσει για να αντιληφθεί η τιμή σταθερή. Ήταν μια πολιτική που προσπάθησε ο πρόεδρος Κλίντον και που απέτυχε. Πανηγυρικά. Και ήταν μια σκέψη που εξέτασε προσεκτικά το κοινοβούλιο και την απέρριψε. Με απόλυτη ψηφοφορία στο σώμα, δις. Ούτε κάνει μια φορά μόνο, γιατί επανήρθε. Ο Στράφος Κλό Τούρμες έπαιξε σημαντικό ρόλο εκεί και άλλοι βέβαια, λέγοντας ότι αυτό ήταν η λύση ενός προβλήματος που δεν υπήρχε. Παρακαλώ Γιάννη λοιπόν προσπαθούσαμε να εργαστούμε ώστε αυτό που έχουμε ήδη να λειτουργήσει καλύτερα, να μην προσπαθήσουμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο. Ευχαριστώ. Έχουμε υπερβεί κάπως το χρόνο ως προς αυτό το σημείο υπάρχουν άλλες τρεις παρεμβάσεις. Θα ήθελα να ζητήσω από τους τρεις συναδέλφους να αποστείλουν γραπτός ε, τις, ερω... τις ερωτήσεις τους για να έχουμε χρόνο για την απάντηση, αν δεν έχετε αντίρρηση. Σας ευχαριστώ πολύ και λυπάμαι πολύ. Θα λάβετε από τον Πρόεδρο όλες τις απαντήσεις γραπτός. Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Δεν έχουμε αρκετό χρόνο για απάντηση των ερωτήσεων, όλων των ερωτήσεων και φυσικά ε, δεν υπάρχουν επακριβείς απαντήσεις, για ορισμένες τουλάχιστον απαντήσεις. Θα πρέπει να πω ότι με εκπλήσει η παρέμβαση του συναδέλφου, του Κλοντ Τούρμες, γιατί το συζήτησα και μαζί σας το θέμα και γνωρίζετε πολύ καλά ότι θα ερχόμουν στην Επιτροπή σας, στην Επιτροπή μας, στην Ήτρε και το συζήτησα και με τους συντονιστές, με συγχωρείτε, των πολιτικών ομάδων. Τους είπα ότι θα παρουσιάσω αυτή την πρωτοβουλία και ένας από αυτούς ήσασταν και εσείς, ε, Κλοντ. Γι' αυτό με εκπλήσει που εκπλήσεστε που βρίσκομαι εδώ. Λυπάμαι, Κλοντ. Uh, μου φαίνεται απίστευτο, απίστευτο πραγματικά. Βεβαίως ε, μπορείτε να μου πείτε ότι ε, πρότεινα κάτι διαφορετικό από αυτό που υπάρχει στην ε, έκθεση, διότι θα ήθελα να σας πω ότι προβάλλω μία πολιτική ιδέα, απαντώντας και σε σένα, Giles, Τσίτσεστερ, γιατί είπε ότι κάνουμε πολλά, το γνωρίζω, το γνωρίζω. Αλλά ξέρεις πόσο δύσκολο είναι. Θυμάσαι τις ε, συζητήσεις μας στο τρίτο ενεργειακό πακέτο. Τι χρειαζόμαστε σήμερα. Χρειαζόμαστε η πολιτική, στη, πολιτική στήριξη για ορισμένες κοινέ ιδέες. Από πού, από τα κράτη-μέλη. Γιατί τίποτα δεν μπορεί να συμβεί χωρίς την υποστήριξη των κρατών μελών έχουμε τις ε, κοινοτικές μας μεθόδους, αλλά σε ζητήματα ζωητικής ε, σημασίας χρειαζόμαστε την υποστήριξη των κρατών μελών και ξέρουμε ότι αυτό είναι ύψης της ε, σημασίας. Τα ανεξάρτητα κράτη-μέλη είναι κυρίαρχα. Γι' αυτό τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε υποστήριξη, Giles, από αυτά. Όλα αυτά γίνονται για μια μεγάλη πολιτική όθηση από, τη, από όλες τις επιτροπές, την έμβη, εμάς, από όλες. Είναι θέματα ύψης της σημασίας και αν μπούμε σε λεπτομέρειες βεβαίως έχουμε πολλαπλή νομοθεσία επιτάπητος. Σας έδωσα και ορισμένα παραδείγματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είναι εύκολο να εφαρμοστούν. Ίσως όχι. Γι' αυτό τουλάχιστον θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τρία σημεία. Τα δίκτυα, ξέρουμε ότι είμαστε ελληματικοί σε αυτό το τομέα. Το δεύτερον, κοινή στρατηγική για την ενέργεια γιατί τα επιτυγχάνουμε όλα χάρη της έρευνας των νέων τεχνολογιών και των ανανεώσιμων. Και τρίτον, υπάρχει μεγάλη ένταση μεταξύ κρατών μελών. Εξαιτία των διαπραγματεύσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται αυτό. Χρειάζεται να έχουμε πληθώρα ερωτήσεων για τον Αμπούκο, το North Stream, το South Stream και όλα τα σχετικά. Όχι, δεν είναι αναγκαίο. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε από κοινού για αυτά τα θέματα. Τρία σημεία είναι πολύ σημαντικά. Μιλάμε για κοινότητα, δηλαδή υποστήριξη ιδεών, τις δικές σας ιδέες, τις δικές μας ιδέες από την Επιτροπή Ήτρε έτσι ώστε να γίνουν πιο κατανοητές τα κράτη-μέλη. Και ζητώ από τους συντονιστές που είναι υπεύθυνοι για τις πολιτικές ομάδες να υποστηρίξουν κάτι τέτοιο. Γιατί παρουσιάστηκε. Το ξέρουν οι συντονιστές ότι σας ρώτησα αν μπορώ να κάνω αυτή την παρουσίαση. Δεν έχω χρόνο, δυστυχώς για να απαντήσω ξεχωριστά σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά η βασική ιδέα ζωτικής σημασίας είναι πολύ ουσιώδης. Είναι η απαρχή νέων ιδεών και θέλουμε τα κράτη-μέλη Ρωτήσατε, ναι εντάξει, επισκέφθηκα 14-15 κράτη-μέλη επίσημα και σε κάθε συζήτηση αυτό ήταν το βασικό μου θέμα. Με πρωθυπουργούς, με υπουργούς και ούτω καθεξής για την κοινότητα. Πώς να αλλάξουμε την προσέγγιση μας σε ενεργειακά ζητήματα. Βεβαίως έγιναν πολιτικές συζητήσεις χωρίς λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες ε, ξεκίνησαν μία ώρα πριν. από τις τρεις και μετά το συζητάμε λεπτομεριακά. Πριν ήταν μια γενική πολιτική ιδέα και οι πρωθυπουργοί σε 15 κράτη μου είπαν ότι είναι πολύ καλή ιδέα γιατί χρειαζόμαστε μία πιο ρωμαλαία Ευρωπαϊκή Ένωση. Κράτη-μέλη και Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ενεργειακά ζητήματα. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι για την υποστήριξή σας. E Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο και ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους που δεν έλαβαν το λόγο. Όπως και να έχουν τα πράγματα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Διαφορετικά δεν θα είχαμε ξεκινήσει μια τόσο σημαντική συζήτηση.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

Madame Πρόεδρε, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία τάση οστρακισμού από τη δική σας πλευρά, λέει ο μιλητής και διακόπτει. Πρέγω, κολέγα. Με συγχωρείτε, δεν άκουγα την διερμηνία, λέει η Πρόεδρος. Merci, Madame la Présidente. Γνωρίζω ότι δεν υπάρχει καμία τάση εξωστρακισμού από, σας πλευρά, από τη δική σας πλευρά, αλλά θα πρέπει να ξαναδούμε τη συνεδρίαση των συντονιστών. Εγώ πάντα ακούω όσα λέγονται και λυπάμαι διότι η ομάδα μας δεν έλαβε το λόγο σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Θα ήθελα στο μέλλον, ακόμα και εάν βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο ε, πλαίσιο συζήτησης, να εξεύρουμε ένα τέτοιο τρόπο συζήτησης έτσι ώστε όλες ε, οι ομάδες να μπορέσουν να εκφραστούν. Διαφορετικά δεν θα είναι δίκαιο, καθόλου δίκαιο. Ε, Πρέπει να σας πω, συνάδελφε, ότι έχετε απόλυτο δίκαιο. Δεν ε, φταίω προσωπικά. Ήταν αδύνατο να ολοκληρώσουμε τον κατάλογο. Αλλά συνειδητοποίησα πραγματικά ότι δεν παρεμβήκατε ως πολιτική ομάδα. Ίσως έπρεπε να ορίσω μία διαφορετική σειρά. Ζητώ συγγνώμη, κάθε πολιτική ομάδα θα πρέπει να μπορεί να παρέμβει. Δυστυχώς ήταν κάτι το εντελώς τυχαίο. Δεν υπήρχε σκοπιμότητα. Καλωσορίζουμε τον Επίτροπο Έτιγκερ. Του ζητούμε συγγνώμη για αυτή την καθυστέρηση οι παρεμβάσεις ήταν ε, μεγάλες. Ελπίζω να είμαστε πιο ε, συγκροτημένοι και συγκρατημένοι στο δεύτερο αυτό θέμα. Ο Επίτροπος θα μας μιλήσει για την έκθεση της Κομισιόν του Απριλίου για το στάδιο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Προγράμματος Ανάκαμψης είναι μια έκθεση που εγκρίνει κάθε χρόνο η Επιτροπή. Πέρα από αυτό το θέμα θα μας μιλήσει για μια πρόταση τροποποίησης του κανονισμού σε σχέση με τη δυνατότητα χρήσης όλων των κονδυλίων και ταμείων που δεν χρησιμοποιήθηκαν ε, μέχρι τώρα. Έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Θα σας παρουσιάσω την πιο πρόσφατη πρότασή μας που εγκρίθηκε μόλις χθε και που αναφέρεται σε πόρους που δεν έχουν ακόμη δαπανηθεί από το Ευρωπαϊκό Διαθετικό Πρόγραμμα για την Ενέργεια. Επιτρέψτε μου πρώτα να σας μιλήσω χθες, ε, για το τι έγινε χθε στο Συμβούλιο Υπουργών Ενεργείας, δηλαδή την συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική του Μέλλοντος το Συμβούλιο συζήτησε ένα είδο απογραφή που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που αποτελεί και τη βάση για την δημόσια διαβούλευση. Τα θέματα που τέθηκαν χθε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργεια αναφέρθηκαν πρώτα σε δομέ, δεύτερον ασφάλεια προμηθειών, τρίτο ανανεώσιμε ενέργειες και τέταρτο αποδοτικότητα τη ενέργεια. Είναι λοιπόν σημαντική ευκαιρία για την Επιτροπή σας να μπορέσει να συμμετάσχει ενεργά στην συζήτηση αυτή για την ενεργειακή στρατηγική, η οποία θα γίνει στο δεύτερο εξάμεινο του τρέχοντος έτους και χαίρομαι ιδιαίτερο που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αφιερώνει το Συμβούλιο που θα γίνει ε, Ιανουάριο και Φεβρουάριο του χρόνου υπό την ηγεσία του κ. Βαν Ρομπόη στο θέμα της ενέργειας όπου θα συζητηθούν εκεί πολλά θέματα και θα αποφασιστούν. Χαίρομαι που αποφασίσατε να συντάξετε έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας και που θα είναι σημαντική για την συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Εγώ βέβαια είμαι στη διάθεσή σας για κάθε είδους συνεργασία. Ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε χθε ήταν η καταστροφή στον κόλπο του Μεξικού. Εγώ εξήγησα τις διάφορες δραστηριότητες που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη συνεργασία με τις πετρελοπαραγωγές εταιρείε στην Ευρώπη και για τις 14 Ιουλίου προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση αυτή με ένα ερωτηματολόγιο για την πρόληψη, για την βελτιστοποίηση των δομών ασφαλείας ώστε να μην συμβεί οτιδήποτε παρόμοιο στην Ευρώπη. Τώρα, επί του θέματος, το Κοινοβούλιο Προέτους ενέκρινε το πρόγραμμα ε, συγκυρίας με 87 προτάσεις οι οποίες αξιολογήθηκαν και από αυτές επελέγησαν 58 για να συγχρηματοδοτηθούν. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία ανέφερε η Πρόεδρό σας από τον Απρίλιο του 2010 για τον, το πρόγραμμα αυτό, δείχνει ότι βρισκόμαστε στον δρόμο. Με 58 λοιπόν project, τα οποία από τα οποία 97% μάλλον τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε 97% δηλαδή 3,8 δις ευρώ θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε. Δηλαδή μεγάλη απορροφητικότητα η οποία προβλέπεται. Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε σήμερα, ένα ποσό 114 εκατομμυρίων ευρώ δεν θα μπορέσει να δαπανηθεί. Για διαφόρους λόγους, και νομικούς και σχεδιασμού δεν είναι υλοποιήσιμα τα σχέδια που έχουν υποβληθεί. Στις 4 Μαΐου λοιπόν εδώ ενώπιόν σας για το πρόγραμμα 2010 σας ανέπτυξα τα σχέδιά μας για τους πόρους αυτούς οι οποίοι δεν είναι δεσμευμένοι. Και είχα συζητήσει και με ορισμένους εκ των βουλευτών σας δημερός προηγουμένως. Χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή μας, πρόταση οδηγίας δηλαδή, που λέει ότι η χρήση αυτών των μη δεσμευμένων πόρων, καθώς επίσης και ενδεχομένως άλλων πόρων που δεν, έχουν, ε, δεν υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν, επιτρέπεται από το EPR δηλαδή. Έχουμε λοιπόν μια καταρχήν έγκριση για να διαθέσουμε τους πόρους διαφορετικά ώστε να μην εκπέσουν μετά την πάροδο των προθεσμιών. Αυτή η πρόταση εφαρμόζει το άρθρο 7 της δήλωσης EEP, δηλαδή μη χρησιμοποιηθέντες πόρους στον τομέα της αποδοτικότητας της ενέργειας και στις ανανεώσιμες ενέργειες. Εκεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά. Εμείς θεωρούμε αυτά τα σημαντικά θέματα αυτά τα θέματα ως σημαντικά, που είναι σημαντικά δηλαδή και για το Κοινοβούλιο και θεωρούμε ότι μπορούν να εφαρμοστούν για την αποδοτικότητα, όπως είπα, της ενέργειας και για ε, έργα ανανεώσιμες ενέργειας, κυρίως σε αστικά κέντρα και σε τοπικές κοινότητες. Αναπτύσσοντας συνέργειες με άλλες δαπάνες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να βελτιστοποιηθεί, να μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητά τους. μέσα στις δυνατότητες που μας ε, επιτρέπουν τα διαφθορτικά ταμεία. Για παράδειγμα, για την βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας σε κτίρια. Η πρόταση αυτή εντάσσεται και μέσα στη στρατηγική του 2020 για την ανάπτυξη και για την απασχόληση. Εμείς προτείνουμε τα έργα αυτά βιώσιμων ενεργειών, για δημόσια κτίρια, για την διασύνδεση παραγωγής ενέργειας και θέρμανσης, για την αποκέντρωση των αναζωσμών ενεργειών, για καθαρή, καθαρές μεταφορές εντός κοινοτήτων κλπ, τον λεγόμενο smart metering, καθώς και την αποδοτική, τον αποδοτικό δημόσιο φωτισμό. Άρα, πρόκειται για ένα ευρύτατο φάσμα χρήσεων, όπου καθίσταται απαραίτητη χρηματοδότηση από πόρους που θα μπορέσουν να έχουν και ένα ρόλο προτύπου. Για να προωθήσουμε πολλά αποκεντρωμένα σχέδια, καλούνται οι τοπικές και κοινωτικές αρχές να υποβάλουν σχέδια, γιατί αυτές θα είναι που θα έχουν και τα πλονεκτήματα. Δηλαδή, ζητούμε συνεργασία των δημάρχων, διότι αυτοί βρίσκονται κοντά στην καθημερινή ζωή του πολίτη και με τον ε, τρόπο αυτό μπορούν να επιτύχουν και τη ταχύτερη δυνατή εφαρμογή. Και με χρηματοδότηση και μέσω τραπεζών και άλλων φορέων που θα παίξουν ρόλο διαμεσολαβητή. Θα ληφθεί υπόψη και μια προσπάθεια, μάλλον και μια προσπάθεια μεγιστοποίησης της βραχυπρόθεσμης απόδοσης των ε, επενδύσεων αυτών για τη δημιουργία και απασχόληση. Θα επικεντρωθεί λοιπόν το μέσον αυτό σε έργα τα οποία μπορούν να αποδώσουν ταχύτατα για την ανάκαμψη, την οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για την αύξηση της ασφάλειας προμήθειας ενέργειας και την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τα κριτήρια του κανονισμού EEPR θα ληφθούν ακόμη περισσότερο υπόψη για τους στόχους του μέσου αυτού. Και κάτι που σας ενδιαφέρει σίγουρα και εσάς, θέλουμε να υπάρξει και μια γεωγραφική εξισορρόπηση των προγραμμάτων και να ληφθεί υπόψη αυτή σε αυτό το νέο πακέτο. Ο χρόνος δεν μας περισσεύει. Η τροποποίηση του κανονισμού πρέπει να εγκριθεί από Συμβούλιο και Κοινοβούλιο πριν από το τέλος του έτους. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λοιπόν συμβαδίζει χρονικά κατευθυνόμενη προς μια πράσινη ανάπτυξη και βιώσιμη. Ελπίζω ότι στην βάση αυτή θα μπορέσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα μαζί με την συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων μερών. Ευχαριστώ για την προσοχή σας σήμερα. Είμαι διαθέσιμος βεβαίως, αν θέλετε και μετά από την συνεδρίαση, για να ε, συνεργαστώ μαζί σας σε οποιοδήποτε επίπεδο και ελπίζω να συνεργαστούμε και στους επόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ας αρχίσουμε την συζήτηση θα παρακαλέσω όλε και όλου να είσαστε το δυνατόν συντομότεροι. Ο κύριος Ρίμπικ πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που προωθείτε τόσο γλίγορα αυτή η μετατροπή το 3 και 98 3,98 δις είναι αυτό για αυτό τον το χρονικό διάστημα και τα 114 εκατομμύρια που απομένουν, τι θα γίνουν ακριβώ. Τα 3,98 δι είναι το συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο μέσα στα πλαίσια των ε, ε, προγραμμάτων που θέλουν να βοηθήσουν για την κρίση. Τα τμήματα του προγράμματο, το ξέρετε, έρευνα, ΕΣΕΣ, ενασιώσιμες πηγές ενέργεια και αποτελεσματική χρήση της και γιατί τότε είχε ε, λεχθεί ότι τα απελευθερώμενα ποσά θα χρησιμοποιηθούν για τι ανανεώσιμε πηγέ και για την αποτελεσματική χρήση. Έχουμε 114 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή Ίσως κάποιο άλλο σχέδιο δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί υπάρχουν νομικά εμπόδια ή γιατί δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση και αυτό ο κανονισμός έχει αυτή τη μορφή. Ίσως μη χρησιμοποιημένοι πορεί, όπως τα 114 εκατομμύρια θα χρησιμοποιηθούν σε σχέδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποτελεσματικής χρήσης ενέργειας. Και για να μην έχουμε μεγάλα κενά χρονικά, εδώ έχουμε κατά νου μικρά σχέδια σε τοπικό επίπεδο, δημόσια ε, αλλά και ιδιωτικά, ούτως ώστε αυτά τα 114 εκατομμύρια θα χρηματοδοτήσουν ένα μεγάλο ρυθμό σχεδίων, ίσως τα περισσότερα κράτη-μέλη μάλιστα. Ευχαριστώ κύριο Χατζημαρκάκη για το λόγο. Δεν θα αναποτείνω στον Επίτροπο να δώσουμε μια ε, συνολική απάντηση. Δεν μπορούμε να απαντάμε σε κάθε, σε κάθε μία ερώτηση. Χατζημακάκης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Εδώ έχουν εγκριθεί περίπου 60 σχέδια. Πολλά από αυτά αφορούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παραδείγματος χάρη τα μεγάλα σχέδια για πάρκα ολικής ενέργειας. Μπορούν αυτά να χρηματοδοτούν Ξέρουμε βέβαια ότι όσο περισσότερα σχέδια ανανεώσιμης ενέργειας προωθούν, τόσο πολύ δυνατότητα αποθήκευσης πρέπει να υπάρχει. Υπάρχουν αυτά. Τα 114 εκατομμύρια μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για αυτού τα σχέδια. Και είπατε, διαστατικά ταμεία και τομεία, ταμεία συνοχής θα πρέπει ακριβώς να ευθυγραμμιστούν περισσότερο και όσον αφορά το δυνατότητα αποθήκευση, τι γίνεται, το έχετε στήσει με του συναδέλφου ιδίω με τον κύριο Χάν, που είναι για τα περιφερειακά υπεύθυνα. Βανιστερόι. Κύριος Βανιστερόι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο γιατί μας διαβίβασε αυτές τις πληροφορίες τόσο σύντομα σε τόσο βραχή χρονικό διάστημα. Φίξαμε ορισμένα ζητήματα τα οποία αποτελούν προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΕΛΚ εδώ και καιρό λέει ότι τα θέματα υποδομής έχουν μεγάλη σημασία, η αιωλική ενέργεια, καθώς και άλλα προγράμματα. Θα πρέπει να εγγυηθούμε αυτά τα προγράμματα σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Θα πρέπει να συζητηθούν γιατί το 97% των κονδυλίων έχει ήδη απορροφηθεί και το Κοινοβούλιο θα ήθελε να γίνει πλήρης χρήση του πακέτου με βάση την ενεργειακή αποδοτικότητα. Μιλάμε για 114 εκατομμύρια αυτό το ποσό, τα 114 εκατομμύρια, τι αφορά. Ίσως θα πρέπει να γίνουν ορισμένες στοχοθετήσεις προτεραιοτήτων, γιατί βλέπουμε τα κράτη-μέλη μεμονωμένα έχουν προωθήσει δράσεις. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν δράσεις, άρα δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνουμε μέτρα που έχουν ήδη προταθεί από τα κράτη-μέλη. Άρα στην πρότασή σας θα πρέπει να δούμε πιο συγκεκριμένα πώς προβλέπετε αυτή την κατανομή. Υπάρχουν χιλιάδες προγράμματα που αναφέρονται. Δεν θα πρέπει να έχουμε απώλειες. Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας. Νομίζω ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πολύ μεγάλη κρίση και όλα όσα είπατε είναι απόλυτα σαφή. Μιλήσατε και για αυτή την διάσκεψη των δημάρχων. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλή σε αυτά τα πλαίσια. to um, Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για αυτή την ανακοίνωση που είναι ιδιαίτερα ε, πρόσδεκτη. Είμαι ε, λίγο απογοητευμένοι, ελάχιστα απογοητευμένοι, διότι αυτό σας το είχαμε πει εξ αρχής. Ως προς το αρχικό, τις αρχικές διαπραγματεύσεις, το σχέδιο ανάκαμψης, προσπαθήσαμε να μπουν χρήματα για την ε, ενεργειακή αποδοτικότητα, γιατί είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει άμεσα και αφορά και την οικονομική όθεση και την απασχόληση. αλλά εν πάση περιπτώσει είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η κατανομή κονδυλίων. Θα πρέπει να υπάρχει μία διασύνδεση με την ε, ΕΤΕ, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα μόχλευσης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και με άλλους φορείς. Αυτό αφορά και την ε, τοπική αυτοδιοίκηση, την ε, διάσκεψη των δημάρχων. Προβλέπετε δυσκολίες από το Συμβούλιο. και πότε μπορεί να επέλθει συμφωνία από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Θα αντιμετωπίσετε δυσκολίες. Κλοντ Τούρμες. Κλοντ Τούρμες. κύριε Πίτροπε, νομίζω ότι η παρουσίασή σας ευθυγραμμίστηκε με αυτό που είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο το φθινόπωρο. Η ερώτησή μου, πολύ σύντομα, είχατε χρόνο χθε στο Συμβούλιο να συζητήσετε με τους υπουργού αυτές τις τροπολογίες. Γιατί το Κοινοβούλιο είναι ενωμένο πίσω σας για την πρόταση αυτή. Και τώρα θα πρέπει να δούμε κατά πόσον το Συμβούλιο έχει την ε, πλειοψηφία για να προχωρήσουμε. La parola collega e-, e... Ο κύριος Μπασίτης και κλείνει ο κατάλογος ομιλητών. Υπάρχουν 5 με 6 παρεμβάσεις. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Και ακτίβια Ιούσου Βίγδομα Πολιτικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο και να σας συγχαρώ για τις αποφάσεις και τις δραστηριότητε σας, ιδίως ε, όσον αφορά την κοινότητα ενέργειας. και για τη δημιουργία ενός κοινοτικού ενεργειακού συστήματος για να βγουν από την απομόνωση οι περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ είναι πολύ σημαντική η αλληλεγγύη. Χωρίς αυτή την αλληλεγγύη δεν θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας. Ε, θεώρησα πολύ θετικό να ακούσω τη θέση σας όσον αφορά την στάση κάποιων τρίτων χωρών στην τροφοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πηγές ενέργειας. Είπατε ότι οι διαπραγματεύσει με τις τρίτες αυτές χώρες θα πρέπει να γίνουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι κρατών μελών. Αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ θετικό. Και ελπίζω ότι θα υπάρχουν τελικά όχι μόνο τα 114 εκατομμύρια, αλλά περισσότεροι πόροι για να χρησιμοποιηθεί αυτό το κοινό κοινοτικό σύστημα ενέργειας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλες τις χώρες που το έχουν ανάγκη. Ο Έντσου, πρίγω. Ο συνάδελφος Έντσου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία για την εξέβρεση αυτών των ε, κονδυλίων υπέρ της ενέργειας, της ανάκαμψης και θα ήθελα να τονίσω ότι επιτελέσατε μεγάλο μέρος των, ε, υποσχέσεών σας στην ε, αρχή της θητείας σας σε σχέση με άλλους επιτρόπους. Θα πρέπει όμως να δούμε και άλλα θέματα που σχετίζονται, παραδείγματος χάρη στην περίπτωση της μόνωσης των κτηρίων, τι προβλέπετε και τι κονδύλια θα δοθούν και σε αυτό το τομέα. La collega Kolaska-Bobinska. κυρία Μπομπίνσκα. Ε, panie Komisarzu, dziękuję bardzo za tak dobry kontakt z Parlamentem. Ευχαριστώ γιατί ήρθατε σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προωθήσατε τόσο καλές σχέσεις. Εάν ανακύψουν διαφορές μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και Συμβουλίου θα ταχθείτε υπέρ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φαντάζομαι, διότι και εμείς είμαστε υπέρ της ενεργειακής αλληλεγγύης. Ε, ως προς τα πάνες του προγράμματος Ναμπούκο, είπατε ότι ίσως ένα τμήμα του προγράμματος ε, δεν θα ολοκληρωθεί. Ίσως δεν θα δαπανηθούν ορισμένα χρήματα. Τι θα γίνει με την περίπτωση του αγωγού Ναμπούκο. Τελειώνουμε με τις παρεμβάσεις και μετά θα απαντήσει ο Επίτροπος, Ευχαριστώ. Μας υποσχεθήκατε να έχουμε στενές σχέσεις και ανταποκριθήκατε σε αυτό. Τώρα που έχετε αναλάβει αυτό το χαρτοφυλάκιο, έχετε την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει αρκετά έναντι των μεγάλων προκλήσεων, διότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και τα κοινοτικά μέσα μιλούν για χρηματοοικονομική υποστήριξη, αλλά εμείς αναμένουμε και ανάκαμψη. Υπάρχει ένα υπόλοιπο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί, αλλά όταν βλέπουμε τη μεγάλη μάζα επενδύσεων στο Γκαλιλαίο, στο Ίτερ, η κυρία Κρούς μας μίλησε για την ευρυζωνικότητα. Πιστεύετε ότι επενδύουμε επαρκώς έτσι ώστε ο πολίτης να έχει εμπιστοσύνη σε μας και σε όλα τα κοινοτικά μέσα. Ε, αν και χρησιμοποιούμε συνεχώς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δηλαδή την προσκολάμε παντού. Και εκεί που πρέπει και εκεί που δεν πρέπει. Είπα ότι πρώτα θα γίνουν όλες οι... θα ακουστούν όλοι και μετά θα δώσει απάντηση ο Επίτροπος. λένε έχεις το λόγο. Κύριε Επίτροπε, εκτιμούμε ιδιαίτερα τον τρόπο διατύπωσης της απόφασης αυτής είναι αποτελεσματική, γρήγορη και όταν μιλάμε για 114 εκατομμύρια ευρώ βεβαίως ε, γίνεται λόγος για συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά και την ΕΤΕ. Άρα τα ποσά είναι υψηλότερα. Εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι έχουμε και υπόλοιπα και αυτό θα το μάθουμε το Δεκέμβριο, κατά τα τέλη Δεκεμβρίου. Αλλά καταβάλλετε κάθε προσπάθεια για να ανακόψετε τη γραφειοκρατία γιατί δώσαμε μεγάλη μάχη στις διαπραγματεύσεις για το χρηματοοικονομικό πακέτο ανάκαμψης, μιλάμε για τις κλιματικές αλλαγές, μιλάμε για απασχολησιμότητα, και τα περισσότερα χρήματα ε, πηγαίνουν σε μακρόπνοα σχέδια που πραγματικά χρειάζονται πολύ χρόνο πριν ε, αποδώσουν. Με την παρούσα κατάσταση στην Ευρώπη χρειαζόμαστε προγράμματα τα οποία να αρχίσουν άμεσα. και εάν χρειαστείτε υποστήριξη για πραγματοποίηση των προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο, μπορείτε να αποτανθείτε και στο Κοινοβούλιο για υποστήριξη, γιατί χρειαζόμαστε γρήγορα σχέδια για την αποδοτικότητα στον τομέα της ενέργειας ήδη από και του χρόνου και όχι το 2020. Κύριε, κολέγα E, e, Ευχαριστώ. Μιλήσατε για 114 εκατομμύρια, μα αυτό είναι μάνα εξ ουρανού. Βάση περιπτώσει δεν είναι πολύ. Ελπίζω κάποια στιγμή να βρούμε χρήματα και από αλλού. Διότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό διακύβευμα, κάτι το οποίο έλυσαν οι Γερμανοί πολύ καλά, όπως και ορισμένες άλλες δυτικές χώρες, δυτικά της Πολωνίας για να το θέσω έτσι. Όσον αφορά τα περιφερειακά ταμεία και πόρους, μόνο ένα 2% πήγε σε θέματα στέγασης στα κτίρια και στην αναβάθμιση των παλαιών κτιρίων, στη μόνωσή τους και ούτω καθεξής. Αυτή η αναβάθμιση των κτιρίων θα αποδώσει άμεσα, γιατί δεν χρειάζονται ε, πρωταρχικά σχέδια εφαρμογής. Θα δημιουργηθούν επίσης και πολλές θέσεις απασχόλησης. Ω προ τα νέα κράτη-μέλη, αυτό είναι η ύψη τη σημασία να το σκεφτείτε για τα νέα κράτη-μέλη. Ζαντό, αλλά παρόλα. Ζαντό. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Για να είμαστε σαφεί, μα λέτε ότι έχουμε ένα 97% του σχεδίου ανάκαμψη το οποίο βρίσκεται σε δαπάνες υποχρεώσεων. Και αυτό το 3% είναι 114 εκατομμύρια, αν κατάλαβα καλά. Δεν μιλάμε για ένα 97% του, των χρημάτων ή των projects που έχουν δεσμευτεί, που έχουν αναλυφθεί. Από ό,τι ξέρω στη Γαλλία υπάρχουν πολύ περισσότερα προγράμματα από αυτά που αναλύθηκαν αυτή η τροποποίηση που προβάλλεται δίνει νέες δυνατότητες, διανοίγει νέες δυνατότητες για το μέλλον. Και εάν δούμε ότι άλλα σχέδια ακυρώνονται, αυτή η τροποποίηση θα αποτελέσει κάτι το σαδεδικασμένο, ας το πούμε έτσι, ως προς την ενεργειακή αποδοτικότητα. Κριστιανέλε. Κριστιανέλε. Κύριε Επίτροπε, οι δομές των κατοικιών ε, συνήθως στην Ευρώπη είναι δύο ειδών. Κατά 60 και 70% των ε, κατοικιών στις πρώην ανατολικές χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού του πρώην ε, βρίσκονται ακόμα στα χέρια του δημοσίου ή των κοινοτήτων και τοπικών αρχών. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι τόσο πολύ οι πόροι, αλλά οι κύκλοι επενδύσεω των ε, ε, διαφόρων αυτών δημοτικών και κοινοτικών εταιριών στέγης. Δεν θα ήταν σωστό αυτοί οι πόροι να χρησιμοποιηθούν κατά κάποιο τρόπο ως μοχλός, ίσως σε συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ώστε να αναπτυχθούν μηχανισμοί χρηματοδότησης που δεν μπορούν να βασιστούν μοναχά σε επιδοτήσεις. Τώρα μάλιστα που υπάρχει και με τη Βασιλεία 2 ο προβληματισμός, για παράδειγμα και στην Ανατολική Γερμανία και σε άλλες ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες, αυτές οι δημοτικές και κοινοτικές εταιρείες έχουν ήδη επενδύσει προπενταετίας, εξακολουθούν και επενδύουν τώρα και μέσω των τραπεζών έχουν τις χέρειες να προχωρήσουν σε μια επόμενη φάση επενδύσεων, διότι οι αναχρηματοδοτήσεις είναι δύσκολο λόγω και των εθνικών δικαίων μισθώσεων που έχουν πάντοτε πολύ μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Επομένως η χρήση των πόρων, των άμεσων πόρων, είναι τελείως ε, διαφορετικές σε άλλες χώρες όπου η κατοικία βρίσκεται κυρίως σε ιδιωτικά χέρια. Γι' αυτό το ερώτημα είναι, κατά τη γνώμη μου, εάν πρέπει να σκεφτεί κανείς εάν οι πόροι που είναι διαθέσιμοι ακόμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να παίξουν το ρόλο ενός μοχλού, όπως είπα, ώστε σε συνδυασμό και με άλλες δυνατότητες επενδύσεων, άλλες δυνατότητες χρηματοδοτήσεων από, για παράδειγμα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, να μπορέσουν να γίνουν χρηματοδοτήσεις και άρα επενδύσεις σε πράγματα που αλλιώς δεν μπορούν να γίνουν. Έκλεισε ο κατάλογος με τους συναδέλφους Ριβαζιέ και Τσικάου. Εντάχει, παρακαλώ. Χαίρομαι διότι τονίζουμε τις ε, προτεραιότητες έτσι ώστε να μειωθούν οι εκπομπές ε, θερμοκηπίου και να τονίσουμε το θέμα της ε, ενεργειακής αποδοτικότητας. Είτε υπάρχουν ε, τέσσερα δις στον ένα ή στον, ένα, στον άλλο τομέα, αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει ενεργειακή αποτελεσματικότητα και αυτό το 20% να μας οδηγήσει σε 100 δις ευρώ. Αυτά τα ευρωπαϊκά ταμεία, η ΕΤΕ, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί περιλαμβάνονται σε όλα αυτά. Ίσως θα πρέπει να δώσουμε ε, κίνητρα και στις ιδιωτικές τράπεζες έτσι ώστε να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή την ε, αλλαγή για τη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Ας δώσουμε λοιπόν κίνητρα στις ιδιωτικές τράπεζες για, την, για τις επενδύσεις ως προς την ενεργειακή αποδοτικότητα. Ένα λεπτό στη συνάδελφο Τσικάου. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, πέρσι η Επιτροπή μας ε, μίλαγε για ένα δις ευρώ το οποίο θα αποδοθεί στην ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων. Μετά είχαμε τον κανονισμό και μπήκε η πρωτοβουλία Smart Cities. Είπαμε δηλαδή ότι δεν έχει δαπανηθεί από το σχέδιο ανάκαμψης θα μπει στο σχέδιο Smart Cities. Ξέρουμε ότι έχουν απομείνει 114 εκατομμυρία για την αποδοτικότητα των κτηρίων, τη μόνωσή τους. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω, ε, ε, συνεργαζόσαστε με τον Επίτροπο Χαν για να ε, προωθήσετε την ενδιάμεση έκθεση το 2010 έτσι ώστε να αυξηθεί η απορρόφηση των κονδυλίων για τη μόνωση των ε, κτηρίων και για τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές προβλέπεται αύξηση έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα 4% ως προς το θέμα της ε, αποδοτικότητας και μόνωσης κτηρίων. Έχετε κατακλειστεί από, τη, από ερωτήσεις, έχετε το λόγο. Κοιτάξτε, φαντάζομαι θα ξεπεράσουμε τα 114 εκατομμύρια. Βέβαια, για αυτές τις ιδέες σας είναι στα γόνα ωκεανό αυτό το χρήματα. Και θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι κάνουμε με τα χρήματα αυτά και ποια είναι η στρατηγική που εκπροσωπούμε και έναντι του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Του επόμενου μήνε τι κάναμε μέχρι στιγμή, αλλάξαμε τον κανονισμό. Γιατί παρατάθη η προθεσμία η υποβολή των αιτήσεων για τα χρήματα αυτά μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Και μετά είπαμε όλα τα χρήματα που απελευθέρονται θα χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματική χρησιμοποίηση ανανεώσιμε πηγέ. Που είναι 114, 80, 30 εκατομμύρια. Παραδείγματο χάνει. Για τον Αμπούκο είμαι περιορισμένη αισιόδοξο είναι σαφές όμως ότι τα χρήματα που προβλέπονται θα χρησιμοποιηθούν εκεί μόνο αν πραγματοποιηθεί ένα μπουκο. Και αυτό που θέλω εγώ είναι τα χρήματα αυτά να μην επιστραφούν στα κράτη-μέλη, αλλά να χρησιμοποιηθούν. Κάθε ένα ευρώ να βρει τη χρήση του. Και γι' αυτό έχουμε μια σταθμισμένη προσέγγιση, δηλαδή ε, παράθεση της προθεσμίας μέχρι το τέλη του έτους και αυτή τη στιγμή διαβλέπονται 114 εκατομμύρια και αν αργότερα έχουμε και άλλα χρήματα που θα απελευθερωθούν, που δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν δηλαδή, θα προσθεθούν στα 114 εκατομμύρια για τους δύο ίδιους στόχους. Και η επεξεργασία στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ε, βοηθήσει να υπάρχει μια προσθέμενη ε, αξία. Ερωτήθηκε επίση όπω έχουμε τι δυνατότητε αποθήκευση ενέργεια. Είμαι σίγουρο ότι το θέμα τη ε, ανανεώσιμη πηγή ενέργεια, ε, υποδομέ και αποθήκευση θα πρέπει από κοινού να εξελιχθούν. Δηλαδή, χωρί αποθήκευση και υποδομή δεν μπορεί να δώσουμε στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια τι κατάλληλε προοπτικέ. Βέβαια, δεν θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε αυτά μέχρι τον Οκτώβριο εγώ ξέρω διάφορα σχέδια, Παραδείγματο ξέρω στο μέλλον αδρυμό, στην πατρίδα μου, όπου υπάρχουν πολλέ αντιδράσει για τη δημιουργία ενό νέου φράγματος. Για σκεφτείτε το, ανησυχούμε ότι όλοι εκείνοι που είναι υπέρμαχοι της ενερώσιμης πηγής ενέργειας προτίθενται να μαχηθούν στο πλευρό μας για την υποδομή, για την αποθήκευση. γιατί θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι θα χρειαστούμε και μια νέα γενιά τεχνολογίας που θα πρέπει τώρα να αναπτυχθεί. Και αυτό δεν γίνεται σε δύο μήνες ή πέντε μήνες. Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα πρόγραμμα ενέργειας αλλά και ένα πρόγραμμα κυρίως ε, συγκυρίας. Και ελπίζουμε ότι το επόμενο έτος θα βγει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την κρίση. Εγώ είμαι φυλεκτικό αλλά ε, τα επίσημα προγνωτικά προβλέπουν ανάπτυξη στα κράτη-μέλη, σε όλα τα κράτη-μέλη για το επόμενο έτο. Θα πρέπει λοιπόν να εθαλύνουμε την ε, συγκυρία. Και αυτό θα πρέπει να βοηθήσει για τι θέσει απασχόληση, για τη βιομηχανία, για του εργαζόμενου, για την προσφορά υπηρεσιών. Και γι' αυτό. Προθεσμία μέχρι τέλη Μαρτίου, οι δύο στόχοι στου οποίου ανέφερα και όποιο ευρώ απελευθερωθεί το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο θα μεταφερθεί και θα προσθεθεί στα 114 εκατομμύρια. Το Συμβούλιο είναι θετικά διακείμενο, το ενημερώνουμε. Ήδη στο σημείο κίνησης αναρωτήθηκαν τα κράτη-μέλη κατά πόσο χρειάζονται εθνικοί πόροι που θα χορηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο. Αυτό ήταν θέμα αρχής που σχετίζεται με το ποιοι είναι οι στόχοι ενέργειας που μπορούν να επιληθούν μόνο ομοιόμορφα στην Ευρώπη. Δίνω την εντύπωση ότι πολλά μπορούν να επιληθούν σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Όχι όλα όμως. Και είχαμε μια επιτυχή συζήτηση με τους υπουργούς ε, ενέργειας της Πολωνίας, Ιστονίας, Βετωνίας και Λιθουανίας για το φυσικό αέριο και για την υποχρέωση όσον αφορά τις υποδομές για την ηλεκτρική ενέργεια. Χωρίς το πρόγραμμά μας δεν θα είχε αποδώσει αυτή η συνάντηση χθε. Μόνο επειδή έχουμε τους σπόρους έχουμε και τη δυνατότητα να προχωρήσουμε. Ολοκλήρωση, λίγη, λιγότερη εξάρτηση από τον Ρώσο εταίρο και ούτω καθεξής. Άμα περάσει η κρίση και περνάμε στη νέα περίοδο ανάπτυξη. τι θα πρέπει να κάνουμε εμεί Έρευνα για την ενέργεια, προώθηση σχεδίων και υποδομέ. Θα καταφέρουμε στον ε, ευρωπαϊκό προπολογισμό τη επόμενη δεκαετία να έχουμε κάποιες ε, κάποια συνεχή κονδύλια για τους στόχους αυτούς που θα πρέπει να πληθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. τίθεται βέβαια και το θέμα με πόση επιτυχία συνεργαζόμαστε εσείς με συναδέλφους σε άλλες ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές, δηλαδή με μας για προπολογισμό. Μετά. Η υπευλήθη ερώτηση θα κάνουμε για την αποτελεσματική χρήση ενέργειας στα παλαιά κτίρια. Θα πρέπει να δούμε τι προωθήσαμε του τελευταίους ε, χρόνους. Automotive, μεταφορές, ε, ε οικονομία τη ενέργειας. Όσον αφορά τα κτίρια, έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατότητα εξοικονομήσεων ενέργειας, αποτελεσματική χρήση της ενέργεια και μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Γι' αυτό συνεργαζόμαστε ένα με τον συνάδελφο Χάν, ο οποίος στο περιφερειακό και η Εθνωτικό του Ταμείο δεν ε, χρησιμοποιεί πάντα όλα τα κονδύλια και ίσως μέσα στα πλαίσια ενός άλλου ε, σχεδίου ε, θα μορφύνουμε το χωριό μας ας πούμε θα χρησιμοποιηθούν και προγράμματα για την εξοικονόμηση ενέργειας από τα παλιά κτίρια. Και γι' αυτό ενδιαφέρομαι πολύ για ένα συνδυασμό των δικών μας στόχων με τους στόχους του συναδέλφου Χάν. Την περασμένη Παρασκευή είχαμε μία διάσκεψη για τις υποδομές στη Μαδρίτη που ξεκίνησε από την Κομισιόν και θα ήθελα να σας πω ότι το θέμα της υποδομής για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό ρίο, κυρίως ηλεκτρική ενέργεια, σε όλα τα κράτη-μέλη, πέρα από αυτά, Μεσόγειος, ε, βο, ε, σκανδιναβικές χώρες, ε, Τουρκία, Ουκρανία, Γεωργία και τους αγωγούς όλο αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα των υποδομών. Μετά θα ακούσετε τον νέο διευθυντή της υπηρεσίας ΕΣΑ, όπου θα πρέπει να υπάρχει ένα συντονισμό των ρυθμιστικών αρχών, όπου θα είναι σαφές ότι θα έχουμε μόνο λίγο από τις δυνατές πρωτοβουλίε στο κοινωνικό επίπεδο και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προωθήσουν όσο μπορούν τις ε, πρωτοβουλίες. Και η Κομισιόν θα έρθει το φθινόπωρο να ξανασυζητήσει τα θέματα αυτά μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο γιατί χρειάστηκε να ε, αντιμετωπίσει μία χιονοστιβάδα ερωτήσεων και σας χαιρετούμε. Qualche minuto per eh, cambiare i nostri relatori. Proseguiamo questo pomeriggio di lavori. Συνεχίζουμε αυτό το απόγευμα, το, με τις απογευματινές εργασίες με εντατικούς ρυθμούς. Όποιος είναι να φύγει στο κάνει τώρα και εντάχει. Proseguiamo i nostri lavori chiedendo appunto... Συνεχίζουμε τις εργασίες μας ελπίζοντας να μας το επιτρέψετε. Καλωσορίζουμε τον δόκτορα Αλμπέρτο Ποτόσνικ που διορίστηκε διευθυντής του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας. Ο οργανισμός υπάρχει εδώ και λίγο καιρό. Ο συνάδελφος Τσίτσεστερ ασχολήθηκε με αυτό το, το θέμα, με αυτή την διασύνδεση. Θα θέλαμε ο Διευθυντής Ποτόσνικ να μας κάνει μία εισήγηση ως προς το πρόγραμμα αυτό, το αρχικό πρόγραμμα, τις προτεραιότητες για τη δραστηριότητα του οργανισμού και μετά θα γίνει μία συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων. Σας καλωσορίζω και έχετε το λόγο. Αγαπητά μέλη, Χαίρομαι και αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ μεταξύ σας, γιατί το Κοινοβούλιο εκπροσωπεί του κατοίκους, τους πολίτες και όταν μιλάμε για αναθεώρηση του τομέα και την, ένα, μια ενιαία αρχή ενέργειας, ξεχνάμε τους καταναλωτές μερικές φορές, άρα θα πρέπει να το έχουμε κατά νου όλοι εμού συμπεριλαμβανομένου. Αναγνωρίζω ότι το Κοινοβούλιο ήταν ένας από τους καλύτερους συμμάχους μας μέσα στα πλαίσια της ε, διαδικασίας κατάρτισης του τρίτου πακέτου για τον οργανισμό. Γι' αυτό χαίρομαι που παρευρίσκομαι εδώ. Όταν με καλέσατε αρχικά, μου ζητήθηκε να καλύψω δύο θέματα. Το πρώτο είναι να σας μιλήσω για την πρόοδο προς τη σύσταση του οργανισμού και το δεύτερο να σας μιλήσω για τις προοπτικές ως προς τα καθήκοντα και τις προτεραιότητες του ε, οργανισμού τους επόμενους μήνες και έτη. Θα ήθελα να ασχοληθώ λοιπόν και με τις δύο πτυχές. Όπως ξέρετε το Διοικητικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Ρύθμισης ορίστηκαν και με διόρισαν διευθυντή και τώρα έχουμε μπει στη φάση σύστασης του οργανισμού. Θα ήθελα να μιλήσω για τρεις πτυχές. Καταρχήν την πρόσληψη προσωπικού, το, τα κτίρια μας και την έδρα μας. Όπως γνωρίζετε, το προσωπικό του οργανισμού θα απαρτίζεται από 42 συν 10 εθνικούς εμπειρογνώμονες. Αυτό προβλέπεται επί του παρόντος και οι πρώτες επτά κενές ε, θέσεις δημοσιεύτηκαν στις αρχές Μαΐου. Τέσσερις επιπρόσθετες δημοσιεύτηκαν χτες. Άρα η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, τουλάχιστον για τον πρώτο πυρήνα του νέου οργανισμού, η φάση αυτή έχει αρχίσει. Μετά αυτό το προσωπικό θα προσλάβει και άλλους οι οποίοι θα ασχοληθούν με την οργάνωση της, ε, του οργανισμού αυτού. Θα αρχίσουμε τη διαδικασία επιλογής νωρίς, ήδη από τον Ιούνιο, ελπίζουμε και φανταζόμαστε ότι θα λήξει η διαδικασία πριν από τον Αύγουστο. Μετά θα δημοσιευθούν και νέες θέσεις αυτό το μήνα και τον επόμενο, έτσι ώστε μέχρι το τέλος του έτους να έχουμε το ίμιση του προσωπικού. Να έχει δηλαδή προχωρήσει αυτή η διαδικασία πρόσληψης. Και άλλοι θα προσληφθούν, οι υπόλοιποι θα προσληφθούν του χρόνου ως προς τον τόπο εργασία μας συνεργάζομαι με τη Σλοβενική κυβέρνηση και με την Κομισιόν για να βρούμε τον κατάλληλο χώρο, το κατάλληλο κτίριο. Έχουμε έξι εναλλακτικές λύσεις ή επιλογές. Ζητήσαμε προτάσεις από τις κυβερνήσεις. Εγώ θα είμαι στη Λιουμπλιάνα την επόμενη εβδομάδα για να ε, διερευνήσω την κατάσταση ως προς τις κτηριακές εγκαταστάσεις και να έρθω σε επαφή και με τη Σλοβενική κυβέρνηση. Η τελική επιλογή θα γίνει τον Αύγουστο και στόχος μας είναι να έχουμε αυτούς τους χώρους έτοιμους μέχρι τη λήξη του έτους. Άρα θα αρχίσουμε τη δραστηριότητά μας στις Βρυξέλλες αλλά μέχρι του χρόνου θα μπορέσουμε να μετακινηθούμε το, να μετακινηθούμε στη Λιουμπλιάνα μέχρι τις 3 Μαρτίου. Ε, ένα σχέδιο στις Σλοβενικές Αρχές το Μάιο. Αυτό είναι το πρώτο θεσμικό όργανο το οποίο έχει έδρα τη Λιουμπλιάνα και κατά την επίσκεψη μου την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουμε άτυπες συζητήσεις. Μετά η έγκριση θα γίνει από το Σλοβενικό Κοινοβούλιο και οι τελικές διαπραγματεύσεις θα λάβουν χώρα αργότερα το καλοκαίρι. Ελπίζω να υπογράψουμε τη συμφωνία για την έδρα το Σεπτέμβριο. Βρισκόμαστε σε μια πρωταρχική φάση εργασιών, προσπαθούμε να επιταχύνουμε τους ρυθμούς μας και ως προς τις προτεραιότητες θα ήθελα να ασχοληθώ με δύο ε, μέρη, τις εσωτερικές προτεραιότητες και τις εξωτερικές. Οι εσωτερικές, όπως φαντάζεστε, καταρχήν είναι να προσλάβω ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού και στη συνέχεια να δημιουργήσουμε μια καλή, ε, καλές συνθήκες εργασίας και μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα εργασίας. Μια άλλη προτεραιότητα είναι να οριστεί ε, μία αρχή δυνατότητας ε, προσφυγών, μία αρχή προσφυγών, έτσι ώστε να μπορέσουν να προσφύγουν οι ενδιαφερόμενοι. Board of Appeal. Και στόχος μας στη συνέχεια είναι να οργανωθούμε στη Λιουμπλιάνα μετά από την αρχική φάση εργασιών στις Βρυξέλλες. Ως προς εξωτερικές προτεραιότητες, στόχος μας είναι να συνεισφέρουμε έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε την ενεργειακή αγορά μέχρι το τέλος της ε, θητείας μου, που είναι πενταετής. Αυτός είναι ο απότερος στόχος. Ως προς ε, πιο άμεσες προτεραιότητες, οι περισσότερες ορίζονται από την ανάπτυξη του τομέα και το, την πρόοδο έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια πιο ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά. Μία από τις βασικές προτεραιότητες είναι να ορίσουμε κατευθυντήριες γραμμές και το πρόγραμμα εργασίας θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο μέχρι το τέλος του μηνός. Τότε θα σας αναφέρουμε και τις προτεραιότητές μας. Υποθέτω ότι θα μιλήσουμε για θέματα ηλεκτρικής ενέργειας, συνδεσιμότητα, ασφάλεια και στο τομέα του φυσικού αερίου θα μιλήσουμε για διαλειτουργικότητα και για συμφωνία ως προς τις τιμές. Με βάση αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές θα, κινηθούμε προς το μέλλον για την κατάρτιση δικτύων. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων ως προς την εργασία των ρυθμιστικών αρχών τους τελευταίους μήνες, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε όλο το υπόβαθρο, όλο το υλικό που χρειαζόμαστε έτσι ώστε να εργαστούμε σωστά. Μία άλλη προτεραιότητα θα είναι να δούμε τα δεκαετή ε, σχέδια ρυθμίσεων. Πιστεύω ότι τα ένσω θα είναι σε θέση να μας παρουσιάσουν το δεκαετές πρόγραμμα μετά το Μάρτιο και εμείς θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε στη συνέχεια. Επίσης, θα έχουμε και το καθεστώς των ένσω εδώ θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε ως οργανισμός. Θα πρέπει να επιτρέψουμε λοιπόν σε αυτούς φορείς να εργαστούν όπως πρέπει. Τέλος, θα ήθελα να υπάρχει μία εποπτική λειτουργία του οργανισμού, δηλαδή να ελέγχουμε τους εμπλεκόμενους φορείς και την κατάσταση της αγοράς. Τώρα, πώς θα πρέπει να λειτουργήσει ο οργανισμός, ποια είναι η προσέγγισή μας. Θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Θα πρέπει να υπάρχει τεχνική προσέγγιση ως προς αυτό, μέσα στα πλαίσια της πολιτικής που είναι ήδη διαθέσιμη και θα συνεισφέρουμε για να ορίσουμε καλύτερα αυτή την πλαισίωση μέσα στα πλαίσια της γνωμοδότησης και συστάσεων προς το Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Επιτροπή, καθώς και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές. Θα προσπαθήσουμε να μείνουμε μακριά από την πολιτική, αλλά πάντα θα συνομιλώ με πολιτικούς, όπως κάνω τώρα στην ε, απαρχή της θητείας μου γιατί η πολιτική είναι η άμεσα ε, εμπλεκόμενη φορείς. Ελπίζω να βασιστείτε στον οργανισμό και σε εμένα για τεχνική βοήθεια και αρρωγή και ελπίζω να συνεργαστούμε ως σύμμαχοι για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς ενέργειας. Ευχαριστούμε τον δόκτορα Ποτόσνικ. Ο κύριος Βιντάλ Κουάντρας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Ποτόσνικ, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την παρέμβασή σας και για τις επεξηγήσεις σας. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στο νέο σας έργο που δεν είναι εύκολο, αλλά πολύ ενδιαφέρον. Αναφερθήκατε σε κάτι το συγκεκριμένο. Ε, ψάχνετε μία κτηριακή εγκατάσταση στη Λιουμπλιάνα. Το Προεδρείο του Κοινοβουλίου ασχολείται με κτηριακά ζητήματα και εγώ ασχολούμαι προσωπικά. Έχουμε εμπειρογνώμονες που ασχολούνται με ακίνητα και με μεγάλη πείρα σε αυτό το τομέα. Άρα, εάν χρειαζόσαστε βοήθεια, διαβουλεύσεις, μια γνωμοδότηση, να γνωρίζετε ότι αυτή η εξαιρετική ομάδα θα μπορούσε να σας ε, βοηθήσει, αν βεβαίως εσείς το επιθυμείτε. Πέραν αυτού, θα ήθελα να επαναλάβω ότι εμείς ταχθήκαμε εξ αρχής υπέρ αυτού του οργανισμού, ο οποίος να διαθέτει αρμοδιότητες έτσι ώστε να μπορέσει να δράσει για μια πραγματική ενία πολιτική στον τομέα της ενέργειας. Ήμασταν ε, υπέρμαχοι αυτού του σχεδίου αυτής της συλλογιστικής και είπαμε εξ αρχής ότι θέλουμε ένα πολύ ε, δυνατό οργανισμό. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε και με το Συμβούλιο βεβαίως. Ίσως το αποτέλεσμα να είναι κάτω από τις προσδοκίες μας, διότι εμείς θέλαμε μια πραγματικά, ένα πραγματικά ρωμαλαίο, έναν εύρωστο οργανισμό, αλλά θα είμαστε αισιόδοξοι. Πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρετε και μέσω εποπτείας, συντονισμού, κατάρτισης εκθέσεων προτάσεων θα ε, τα καταφέρετε αν χρησιμοποιήσετε σωστά όλα αυτά τα εργαλεία. Θα πρέπει να έχετε αποφασιστικό ρόλο και εδώ αναφέρομαι στις ε, διασυνοριακές υποδομές. Ας υποθέσουμε θεωρητικά ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο διασυνδεσιμότητας. Και οι χώρες, οι εμπλεκόμενες χώρες δεν συμφωνούν ως προς αυτή τη διασύνδεση, μία μορφή διασύνδεσης. Πείτε μου λοιπόν σας παρακαλώ, ποιος θα είναι ο ρόλος του οργανισμού σε αυτή την ε, υποθετική περίπτωση. πώς θα μπορέσει να συνεισφέρει ο οργανισμός για να ε, δημιουργήσει, για να φτάσει σε μια απεμπλοκή της κατάστασης, στην τελικαστήγιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστούμε κύριε Ποτόσνικ. Να σας καλωσορίσω και εγώ. Εξ ονόματος ε, της ομάδας μου είμαι συντονίστρια. Βρισκόμαστε σε μια στιγμή όπου θα πρέπει να τεθούν σε λειτουργία ε, αυτοί οι δύο φορείς και ο δικός σας ο οργανισμός, τον οποίο εγκρίναμε κατά την προηγούμενη θητεία. Μιλώ για τις Ευρωπαϊκές Ρυθμιστικές Αρχές, το ΑΜΠΕΡΙΚ για την ηλεκτρονική επικοινωνία και το δικό σας οργανισμό. Χτες η Επίτροπος Κρούς μας είπε ότι τελικά το Συμβούλιο χτες το πρωί ενέκρινε την ε, έδρα του άλλου οργανισμού που θα είναι η Ρήγα. Άρα και οι δύο οργανισμοί θα αρχίσουν να λειτουργούν παράλληλα τόσο και ο άλλος οργανισμός, ο Μπέρεκ και ο δικός σας οργανισμός θα αντιμετωπίσετε ορισμένα παρόμοια προβλήματα. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι εξαρτάστε από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Πολλές φορές οι εθνικοί ρυθμιστές είναι πηγή προβλημάτων για τον οργανισμό. Στην περίπτωση του ενεργειακού τομέα υπάρχει πρόβλημα τέτοιου είδους, το οποίο δεσπόζει και θα αποτελούσε ενδεχομένως πρόσκομα στην ομαλή λειτουργία του οργανισμού. Πώς θα μπορούσε να επιληθεί κάτι τέτοιο. Γιατί ε, πρόκειται για υπαρκτό πρόβλημα, τουλάχιστον σε ορισμένα ε, προβλήματα. Η κυρία Ποδηματά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δόκτωρα Ποτότσινγκ, και επιστρέψτε μου να σας συγχαρώ και εγώ από την πλευρά μου και να σας ευχηθώ καλή θητεία. Ε, γνωρίζετε ασφαλώς ότι αναλαμβάνετε καθήκοντα σε μια ε, ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή. Όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, το Κοινοβούλιο θα προτιμούσε έναν ακόμα περισσότερο αναβαθμισμένο και ε, ενισχυμένο ρόλο για τον Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Οργανισμό Ενέργειας, αλλά σε κάθε περίπτωση ε, αναλαμβάνεται καθήκοντα σε μια συγκυρία κατά την οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή η συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία θέτει τις βάσεις για μια κοινή ενεργειακή πολιτική. Πρόσφατα είχαμε και την παρουσίαση της πρωτοβουλίας του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ενεργειακής κοινότητας. Όλα αυτά συγκλίνουν στο ότι η ενέργεια και στις τρεις τις πτυχές και σε ό,τι αφορά την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας αλλά και την ικανοποίηση των ενεργειακών και κλιματικών στόχων της Ένωσης αποκτά ε, καταλητικό ρόλο και πολύ μεγάλη σημασία για το επόμενο διάστημα. Επιτρέψτε μου δύο ερωτήματα να σας θέσω. Το πρώτο αφορά στις ε, αναφορές σας για, την, ε, για το δεκαετή σχεδιασμό σε ό,τι αφορά τα δίκτυα. Είναι ένα θέμα που ετέθηκε από τον συνάδελφο Βίνταλ Κουάντρας πριν. Το ερώτημα είναι τι πρωτοβουλίες και τι δυνατότητες έχει ο οργανισμός ε, για να υπερβεί τον κατακαιρματισμό και την αποσπασματική προσέγγιση που υπάρχει σήμερα στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό για την ε, ανάπτυξη των ε, δικτύων ενέργειας και σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο και σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό στο μείζον θέμα των διασυνδέσεων. Και το δεύτερο ερώτημα αφορά στην, ε, στους Ευρωπαίους καταναλωτές, αναφερθήκατε κι εσείς πριν, συχνά τίνουμε να ξεχνάμε τους Ευρωπαίους καταναλωτές που πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της ε, προσοχής μας. Στο πλαίσιο των συζητήσεων που είχαμε εμείς ε, για το τρίτο ενεργειακό πακέτο, συμφωνήσαμε σε μια χάρτα δικαιωμάτων των καταναλωτών ενέργειας, η οποία ενσωματώθηκε ως παράρτημα στις αποφάσεις μας για το τρίτο ενεργειακό πακέτο. Είναι ένα θέμα που αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία, διότι υπάρχουν ανησυχητικά μηνύματα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας σε πολλές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και μάλιστα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ε, εάν και ποιες πρωτοβουλίες σκοπεύετε ε, να αναλάβετε ακριβώς για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των Ευρωπαίων καταναλωτών ε, ε, ενέργειας και να συγκρατηθούν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. La parola alla collega Maglia Sartori. Grazie Presidente. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω τον νέο διευθυντή του Οργανισμού Συνεργασίας Ρυθμικών Αρχών. Τον ευχαριστώ γιατί μας έκανε αυτή την παρουσίαση γνωστοποιώντας προβλήματα τα οποία είναι δύσβατα όπως όλοι γνωρίζουμε, ιδιαίτερα στη, ως προς την αρχή νέων ε, δραστηριοτήτων. Ελπίζουμε να μπορέσετε να κινηθείτε εντάχει με βάση το πρωταρχικό σας μέλημα, το οποίο και εμείς βιώσαμε με τη συζήτηση που έγινε. Όταν μιλάμε για συμφέροντα καταναλωτών, in primis, μας ενδιαφέρει να ε, ε, μάθουμε πώς εν ευθέτω χρόνο μπορούμε να φτάσουμε σε μία εναρμόνιση μεταξύ κρατών μελών. Αυτό είναι το πρωταρχικό μας μέλημα. Γιατί μία ενιαία, για να υπάρξει μία ενιαία αγορά ενέργειας θα πρέπει να υπάρχουν εναρμονισμένοι κανόνες όπου ο οργανισμός σας θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Οπωσδήποτε χρειάζονται νέοι κανόνες για να συνεργαστείτε με το Συμβούλιο και με μας. Δεν πρόκειται για μία τάχιστη διαδικασία. γιατί έχετε να αντιμετωπίσετε και μία πληθώρα γνωμοδοτήσεων και συστάσεων. Πρώτον, για να φτάσω στις ερωτήσεις μου, ποια είναι η προθεσμία, ποιες προθεσμίες προβλέπονται σε σχέση με την ενδυνάμει εναρμόνιση της αγοράς ενέργειας στα κράτη-μέλη. Και δεύτερον, πώς προτίθεστε να εργαστείτε σε σχέση με τις δυσκολίες που ενδεχομένως ανακύψουν μεταξύ κρατών. τι θα γίνει ως προς ε, ε, αποκλίνοντα συμφέροντα, ως προς τον ενεργειακό εφοδιασμό. Γιατί αυτό είναι ένα από τα ζωτικά ζητήματα που μας ε, απασχολούν αυτούς τους μήνες. Ο κύριος Τούρμες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στον κύριο Ποτότσνη για την ανάληψη αυτών των σημαντικών καθηκόντων. Νομίζω ότι είναι ο πρώτος διευθυντής τέτοιου ιδρύματος, τέτοιου οργανισμού. Και ε, πάντα ο πρώτος πρόεδρος τέτοιου οργανισμού μπορεί να διαμορφώσει τον οργανισμό με κάποιο τρόπο. Το κοινοβούλιο, όπως είπε και ο, και ο Αλέχο Βιδαρκουάδρας, θα ζητήσει, άλλωστε το, το Συμβούλιο Υπουργών έχει προχωρήσει ε, έχει προβάλει ε, διάφορα τρίκ ήδη από τον, τότε που δεν υπήρχε καν η ενιαία αγορά, ούτε κανεί είχε σκεφτεί ε, να κάνει κάτι τέτοιο. Πάντως προσπάθησαν με κάθε τρόπο να αναχαιτήσουν την προσπάθεια αυτή και να μας κόψουν, να ανακόψουν από κάτι που θέλαμε να κάνουμε, που ήταν αυτός ο οργανισμός δηλαδή. Πάντως, σήμερα το πρωί αποφασίσαμε μεταξύ των συντονιστών, δεν θα το γνωρίζετε ακόμη, ότι προτιθέμεθα να ιδρύσουμε μια ομάδα μελών της παρούσας Επιτροπής μια ομάδα λοιπόν ευρωβουλευτών οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξετάζουν τακτικά και να παρακολουθούν τις δραστηριότητές σας. Μία συγκεκριμένη ερώτηση για σήμερα. Έχουμε 12 εταιρείες ενέργειας στην Ευρώπη που κυριαρχούν στο 95% της αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος και αερίου. Αυτές οι επιχειρήσεις. Δεν μπορούμε να τις ρυθμίσουμε αυτές με 27 εθνικούς νομοθέτες. Τι ιδέα λοιπόν έχετε, πώς θα μπορούσε λοιπόν ο οργανισμός σας να συμβάλλει στο να αρθεί στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο η προσέγγιση και η σκέψη, η κοινή σκέψη των 27 αυτών εθνικών νομοθετών όταν πρόκειται για θέμα ρύθμισης της ε, ευρωπαϊκής αγοράς αερίου και ρεύματος. Ο κύριος Ρίμπικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ νομίζω ότι είναι καλό που δημιουργήθηκε ένα νέο πλαίσιο. Συγχαίρω για την ανάληψη των δραστηριοτήτων του τον κύριο Ποτόσνικ. Πρόκειται περί του ότι είναι νέος οργανισμός, ο οποίος θα καταστήσει δυνατή την πρόσβαση εκάστου φορέως, εθνικού φορέως δηλαδή, στις άλλες 26 αγορές, ώστε να μπορούν οι φορείς αυτοί να δραστηριοποιούνται και στις υπόλοιπες εθνικές αγορές. Ένα θέμα που τίθεται λοιπόν είναι το θέμα των διαδικασιών εγκρίσεων. Πρώτη ερώτηση. Έχετε σκοπό να αναζητήσετε τις best practices στις διαδικασίες εγκρίσεων και να κάνετε προτάσεις για μια νομοθετική ρύθμιση στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεύτερη ερώτηση. Σήμερα το πρωί μεταξύ των συντονιστών αποφασίσαμε σε ό,τι αφορά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ε, αντισταθμίσεις που δίνονται σε τρίτα δίκτυα να τα συζητήσουμε. Ήδη έχουμε κάνει πρώτα μια συζήτηση στο Κοινοβουλίο με ψηφοφορία η οποία ήταν με πολύ περιορισμένη προψηφία. Γνωρίζετε ότι για τις μεταφορές αποδόσεων σε άλλα δίκτυα προβλέπονται μοναχά 100 εκατομμύρια περίπου ευρώ. Η ΕΣΑ θα ανασχοληθεί με την ε, απόφαση αυτή της Κομισιόν και πιστεύετε ότι μέσα σε δύο χρόνια θα μπορεί να γίνει ένα assessment στα πλαίσια αυτά και ότι θα μπορεί να κατατεθεί επιτάπητος ώστε αυτή ε, η συζήτηση μεταξύ των ISO να μπορέσει να λυθεί. Ευχαριστώ, Οντί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω και εγώ με τους συναδέλφους μου στην έκφραση συγχαρητηρίων προς τον ε, νέο πρόεδρο, προς τον νέο μάλλον. Σύντομη ερώτηση. Επίπεδο διαφάνειας αποφάσεων του οργανισμού εξαρτάται από τη δική σας δύναμη, από ποσάς να θέσετε υπόψη των βουλευτών και μέσω αυτών του κοινού τις αποφάσεις σας, τις μελέτες κτλ. Ή έχει ήδη καθοριστεί αυτό από τον κανονισμό σας. Γνωρίζετε ότι είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε θέματα διαφάνειας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα επίπεδα. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ποτνότσνικ, θα ήθελα καταρχήν και εγώ να τον ευχαριστήσω και να συμφωνήσω με όλα όσα προελέχθησαν ως προς την διαφάνεια στις πληροφορίες γιατί εμείς συνεισφέρουμε αποτελεσματικά στη δημιουργία οργανισμών και μετά δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Ελπίζω λοιπόν να έχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα ανταλλαγή απόψε. Θα ήθελα να πω ότι το Κοινοβούλιο θα επιθυμούσε και στον τομέα των ε, τηλεπικοινωνιών και σε αυτό το τομέα των ρυθμιστικών αρχών να έχει μια μεγαλύτερη και πιο εύρωστη ευρωπαϊκή αγορά. Βεβαίω να μην έχουμε πολύ υψηλέ προσδοκίες σε σχέση με τις ε, πραγματικές αρμοδιότητε. Αν μπορούσα να κάνω μια σύσταση λοιπόν, θα έλεγα να έχουμε έναν πολύ καλό βαθμό συνεργασίας με βάση το καθεστώς του οργανισμού. Γιατί εμείς επιθυμούμε την εναρμόνιση, την ολοκλήρωση μιας ενίας αγοράς. Αλλά πάντα στο μέτρο του δυνατού. με βάση το τελικό κείμενο ως, όπως προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Θα θέλαμε ο οργανισμός να είναι ιδιαίτερα δυνατός και να ανταποκριθεί στο έργο Το Έχετε το λόγο. Ο Διευθυντής, σας ευχαριστώ για τις ευχές σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα αγγλικά θα είναι ευκολότερο για να κατανοήσετε όλοι. Βίταλ Κουάδρας. Ευχαριστώ για την προσφορά υποστήριξης ε, σε πρακτικά θέματα. Θα γνωρίζω περισσότερα μετά την, ε, μετά την επόμενη συγγνώμη, Τρίτη, όπου θα βρεθώ εκεί, θα είμαι επιτόπου δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι δηλαδή ε, να βρεθεί το κατάλληλο ακίνητο και ίσως να προσφύγω στην προσφορά σας. Ας έρθουμε ε, σε πιο ε, ε, ενδιαφέροντα θέματα. Νομίζω ότι το θέμα των διασυνδέσεων ασφαλώς είναι πολύ επίκαιρο. Ο οργανισμός, ο οργανισμός δεν έχει αποφασιστική αρμοδιότητα. Έχει όμως ένα ηθικό ρόλο πειθούς και σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση, θα έρθω εδώ και στην ερώτηση που έγινε. Θα έρθω σε λίγο σε αυτήν. Σχετικά με το τι μπορεί να κάνει ο οργανισμός για την ολοκλήρωση. Μπορεί να κάνει διάφορα πράγματα ο οργανισμός. Μπορεί πρώτα θα ε, εκδίδει γνωμοδοτήσεις για τον δεκαετή σχεδιασμό των δικτύων. Η γνωμοδότηση θα βασίζεται στην καταλληλότητα και επάρκεια των δικτύων για την υποστήριξη της ενιαίας αγοράς. Εάν ο οργανισμός θεωρήσει ότι τα σχέδια είναι περιοριστικά του ανταγωνισμού ή περιοριστικά της δυνατότητας ανάπτυξης των δικτύων μεταξύ των διαφόρων χωρών μελών, τότε ασφαλώς θα βγούμε και θα το πούμε. Αυτός, εν πάση περιπτώσει, θα είναι ο ρόλος του οργανισμού. Επίσης, ρόλο θα έχουμε την προσπάθεια επίλυση του θέματος της χρήσης των τρέχουσών ικανοτήτων. Θα έχουμε πάλι συμβουλευτική αρμοδιότητα, θα μπορούμε να εκδίδουμε γνωμοδοτήσεις, από την άλλη μεριά μπορούμε να παρέμβουμε εφόσον δούμε ότι οι εθνικοί νομοθέτες δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε ό,τι αφορά την ε, διαχείριση τη ικανότητα διασύνδεση μεταξύ των χωρών μελών ή αν αποφασίσουν από κοινού οι εθνικοί νομοθέτε να παραπέψουν το θέμα στον οργανισμό τότε έχουμε ε, αποφασιστική αρμοδιότητα η οποία είναι δεσμευτική ε, για τους φορείς. Άρα, ο οργανισμός δεν θα απόσχει από το να σηματοδοτήσει όταν θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα με τις διασυνδέσεις που ε, θα, θεωρεί ότι πρέπει να επιληθεί με τρόπο οικονομικά βιώσιμα. βιώσιμο. Συγγνώμη. Τώρα για την κυρία Δικαστήριο για την ε, διασύνδεση των νομοθετών. Το τρίτο, η τρίτη δέσμη μέτρων ενέργειας, αφού το δεύτερο ζητούσε από τους ρυθμιστές να είναι ανεξάρτητοι από την βιομηχανία, από τον κλάδο, το τρίτο λέει ότι πρέπει να είναι οι ρυθμιστές ανεξάρτητοι από την διοίκηση. Αυτή τη στιγμή εφαρμοστεί λοιπόν το τρίτο πακέτο, θα δούμε και πώς θα εφαρμοστεί στις διάφορες χώρες μέλη, αλλά τα στάνταρτ της ε, ανεξαρτησίας των εθνικών ρυθμιστών θα πρέπει να είναι πολύ υψηλότερα από αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι βέβαια πάντοτε ξεκάθαρε οι λύσει, διότι πάντοτε υπάρχει η δυνατότητα της διοίκηση να εγκρίνει επίσημα ορισμένες από τις δράσεις των ρυθμιστών. Ελπίζουμε πάντως του χρόνου να έχουμε πιο ανεξάρτητους ρυθμιστές και αυτό βέβαια θα συμβάλλει και στο έργο του οργανισμού, γιατί είναι πολύ ευκολότερο να συνεργαστεί κανεί με ανεξάρτητους ρυθμιστές παρά με ρυθμιστές οι οποίε έχουν ήδη πολιτική εντολή από τις χώρε μέλη. Το θέμα τώρα των καταναλωτών ενέργειας της κυρίας Ποδηματά, εγώ συμφωνώ ε, μαζί σας, όπως είπα και εγώ είναι μεγίστη σημασία το θέμα. Θεωρώ ότι ο οργανισμός θα μπορέσει να βοηθήσει τους καταναλωτές με δύο τρόπους. Αφενός θα προσπαθήσουμε να προαγάγουμε τον ανταγωνισμό και μια ενιαία αγορά. Ο ανταγωνισμός θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των τιμών, τουλάχιστον απέναντι στο επίπεδο όπου θα αναμέναμε να φτάσουν. Στην αρχή μας λέγανε πού είναι η μειώση των τιμών όταν αρχίσαμε με τους ανεξάρτητους ρυθμιστές και την απελευθέρωση. Η ε, σύγκριση θα γίνεται με το επίπεδο των τιμών που θα έφταναν αν δεν υπήρχε το πακέτο. Μεγαλύτερος ανταγωνισμός λοιπόν θα σημάνει και περισσότερα δικαιώματα υπέρ των καταναλωτών, καλύτερο ηλεκτρικό ρεύμα δηλαδή, δηλαδή με καλύτερου όρου. Ο, ο, ο οργανισμό έχει ως έναν από του σημαντικότερου στόχους να προωθήσει την ενιαία αγορά. Είπα ήδη τους κώδικες των δικτύων που για πρώτη φορά θα είναι δεσμευτικοί σε ολόκληρο σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης και για θέματα δηλαδή όπως επέκτασης δικτύων και άλλων που θα βρίσκονται στην καρδιά της ενιαίας αγοράς. Και ο οργανισμός θα έχει και ευθύνη για την παρακολουθήση, το monitoring δηλαδή, των λιανικών τιμών. Ο οργανισμός λοιπόν θα παρακολουθεί πώς διαμορφώνονται οι τιμές λιανικής ε, στις χώρες μέλη και αν διαπιστώνονται κάποιες ανομαλίες και αν διαπιστώνονται κάποιες ανομαλίες αυτό θα αποτελεί αντικείμενο συστάσεως από πλευρά του οργανισμού ή εν πάση περιπτώσει θα θέτει το θέμα υπόψη των εθνικών ρυθμιστών του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Για την κυρία Σαρτόρη που έδειξε ενδιαφέρον για την εναρμόνιση και για τις προθεσμίες που υπάρχουν. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι από του να παραμείνουμε μοναχά σε ένα επίπεδο εναρμόνισης, να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε, να εντάξουμε τις αγορές. Υπάρχουν ορισμένε προτεραιότητε που ε, αναμένουν να δημοσιευθούν από τον οργανισμό στους πρώτους μήνες της λειτουργίας του όπως είπα, πολλή εργογή έχει γίνει και γίνεται και τώρα από τους ρυθμιστές, ώστε ο οργανισμός θα μπορέσει να προχωρήσει με μεγαλύτερη ταχύτητα. Αυτή τη στιγμή αρχίζει να λειτουργεί. Για τους τομείς που ανέφερα, σε αυτές θα, δοθούν, θα δοθεί ύψιστη προτεραιότητα στις framework guidelines, οι οποίες θα υποβληθούν στο κοινοβούλιο για να εγκριθούν αναμένω αυτές οι αρχικές ε, κατευθύνες γραμμές πλαίσια θα υπάρχουν μέχρι το αργότερο τα τέλη του επόμενου έτους. Αλλά αυτές οι guidelines είναι το πρώτο βήμα σε μια διαδικασία η οποία θα καταλήξει εν τέλει στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των ε, κωδίκων δικτύων. Θα αναπτυχθούν λοιπόν πρώτα αυτές ε, οι κατευθύνες γραμμές, μετά οι κώδικες ο οργανισμό θα παρακολουθεί ότι οι κώδικες συμμορφώνονται με τι κατευθυντικέ γραμμέ μετά θα περάσουμε στην επιτροπολογία και στον έλεγχο, σκρούτινη και αυτά θα είναι τα υπόλοιπα βήματα, τα οποία όμω άλλα βήματα αυτά είναι κάπω εκτό ελέγχου του οργανισμού. Αν προσπαθήσουμε να κάνουμε την δουλειά μα δηλαδή σχετικά γρήγορα, ελπίζουμε ότι και τα άλλα βήματα θα ακολουθήσουν με την ίδια ταχύτητα. Σε ό,τι αφορά την σχέση μεταξύ των διαφόρων χωρών, όπως είπα πριν, ο οργανισμός έχει την ευθύνη να παρεμβαίνει ε, όταν οι ρυθμιστές των διαφόρων χωρομερών συμφωνούν ότι την απόφαση θα λάβει ο οργανισμός ή αν εν τέλει δεν συμφωνούν οι ρυθμιστές μεταξύ τους και αν μετά πάροδο 6 ή 12 μηνών, αναλόγως της περιπτώσεως, την απόφαση αναλαμβάνει πλέον να λάβει ο οργανισμός. Άρα ο οργανισμός θα έχει αρμοδιότητες και ευθύνε να παρεμβαίνει όταν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των διαφόρων ρυθμιστών. Τούρμες. Ναι, είμαστε καλύτερα τώρα που έχουμε 12 χώρες μέλη από ότι παλαιά που υπήρχε μονάχα μία. Δεν ε, σημαίνει απαραίτητα τώρα ότι πρέπει να γίνει ρύθμιση ή εν πάση περιπτώσει η ρύθμιση πρέπει να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα στις αγορές και ότι υπάρχει ανταγωνισμός, δηλαδή διαγωνιστική αγορά σε ολόκληρη την Ένωση. Και μετά ο ανταγωνισμο κατά πάσα πιθανότητα θα διασφαλίσει ώστε οι οι ε, επιχειρήσεις αυτές, οι εταιρείε αυτές να μην μπορούν να καταχρώνται τις δεσπόζουσες θέσεις τους. Όσο μεγαλύτερη αγορά, όσο μεγαλύτερη ενιαία αγορά, τόσο μεγαλύτερος ανταγωνισμός μεταξύ μεγάλων εθνικών επιχειρήσεων ή, εθνικο, ή, περιφερειακών επιχειρήσεων που δεν είναι τόσο μεγάλες αν συγκριθούν με το ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Αυτός είναι ο στόχος, νομίζω, της ολοκλήρωσης της αγοράς σε πρώτο βαθμό. Ασφαλώς ο οργανισμό θα παρακολουθεί, θα παρακολουθεί την εξέλιξη τη αγορά και εάν υπάρχουν προβλήματα, όπως είπα και πριν, θα είμαστε βέβαια έτοιμοι να τα ε, εντοπίσουμε, να τα ε, καταστήσουμε γνωστά και προς εσάς και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Ρούμπικ, με ρωτήσατε για την διαδικασία με την οποία η ΕΝΣΑ θα εγκρίνει και αν θα ε, ακολουθούμε τις βέλτιστες πρακτικές. Θα έχουμε την δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε την, την εμπειρία μάλλον όλων των ρυθμιστών στην Ευρώπη. Υπάρχουν θετικέ θετικές εμπειρίες. Εγώ έχω συνεργαστεί με τους Ιταλούς ρυθμιστές και με την Σχολή της Φλωρεντίας για πολλά χρόνια, όπου είχαμε κάνει εργαστήρια ανταλλαγής απόψεων πολλών ρυθμιστών και νομίζω ότι μπορεί κανείς να διδαχθεί πολλά από τους εθνικούς ρυθμιστές σε ό,τι αφορά την χρήση βέλτιστων πρακτικών. Και ελπίζω ότι το προσωπικό της ΕΝΣΑ θα μεταφέρει αυτήν την ε, ε, νοοτροπία της χρήσης βέλτιστων πρακτικών, αυτήν την κουλτούρα των εισαγωγικών από τις διάφορες γωνίες της Ευρώπης. Ο μηχανισμός ITC, Inter-Tier Compensation, είναι ένα από τα θέματα που σύμφωνα με τον 714 κανονισμό μπορεί να ρυθμιστεί μέσω κατευθείαν γραμμών πλαισίων. Αυτό ε, θα έχει ήδη γίνει. Βέβαια, ο οργανισμός θα παρακολουθεί πώς λειτουργεί, τι αποδίδει το σύστημα αυτό και αναλόγως θα αναφερόμαστε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Ότι διαφάνεια. Ο οργανισμός έχει εντολή να διαβουλεύεται εκτεταμένα για οτιδήποτε πράττει. Πριν λοιπόν ληφθεί η αδίποτε απόφαση θα προηγείται περίοδος διαβουλεύσεων και πάλι εδώ θα φροντίσω να εκμεταλλευτώ τις βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες των ρυθμιστών. Η ΕΡΓΕΓ έχει αναπτύξει ε, μια ολόκληρη πολιτισμό διαβουλεύσεων. Ε, σε ό,τι αφορά την διαφάνεια, όλες οι αποφάσεις του οργανισμού θα δημοσιεύονται μαζί με το υποστηρικτικό υλικό, εκτός από το υλικό εκείνο που θα κριθεί απόρριτο. Εν τέλει δε, κυρία Πρόεδρε, γνωρίζω ότι υπάρχουν υψηλέ προσδοκίες και εγώ έχω υψηλέ προσδοκίες και για τον εαυτό μου αλλά και για το προσωπικό με το οποίο συνεργαστώ στον οργανισμό και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ψηλές αυτές προσδοκίες. Ευχαριστώ. E σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχόμαστε ε, να μπορέσετε να ανταποκριθείτε στις εργασίες σας και σας ευχαριστούμε και πάλι. Ευχαριστώ Sí. Proseguiamo i nostri lavori chiedendo ai nostri ospiti di accomodare. Θα θέλαμε να ζητήσουμε από τους καλεσμένους μας να καθίσουν. Diamo il benvenuto. Sì, prego. Can I put a, a question of method at the beginning? I think this is uh, μια διαδικαστική ερώτηση πρώτα. Μας μένουν 45 λεπτά. Μπορούμε να προχωρήσουμε εις τρόπον ώστε να ακούνε τρεις ερωτήσεις και μετά να απαντούν. Όχι 10 και 12 ερωτήσεις, γιατί μετά οι απαντήσεις δεν μπορούν να είναι ακριβείς. Τρεις ερωτήσεις και μετά απάντηση. Αυτό θα προσφέρει περισσότερο δυναμισμό ε, στην διαδικασία έρωτα αποκρίσεων. Συμφωνώ μαζί σας, ναι, ναι, λέει η ε, Καλώς ήρθατε στους προσκεκρισμένους μας. Κουιντάνα Τρίας, Διευθυντής Ενέργειας της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας, Φραντς Μπρίσκο, της Fusion for Energy, που πρόσφατα διορίστηκε στην αρχές του έτους. Πριν σας δώσω τον λόγο, σας ορίζω. Ζητώ συγγνώμη που έχει εγγραφεί με κάποια καθυστέρηση το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Και ε, θα συζητήσουμε τις ε, διάφορες εξελίξεις στα προγράμματα εργασίας στα πλαίσια της πυρηνικής σύνδεξης για την παραγωγή ενέργειας και θα σας παρακαλέσω να έρθετε και σε θέματα χρηματοδότησης. Διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι και να δούμε εάν φαίνεται επαρκής η χρηματοδότηση ή όχι. Επίσης, να πείτε καθαρά και το πώς θα προχωρήσουν οι διάφορες φάσεις δημιουργίας του ε, project αυτού. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας της Επιτροπής. Ευχαριστώ και καλό σας απόγευμα. Η συμφωνία ITER υπογράφηκε από την Ευρατών και άλλα έξι μέρη, Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, Κορέα, Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες το 2006. Η συμφωνία βασίστηκε σε υπολογισμό κόστους του 2001, άρχισε να λειτουργεί το 2007 και μετά από εκτίμηση ενός ανεξάρτητου πάνελ που προβλέπει διπλασιασμό των ε, εκτιμήσεων αυτών με τον στόχο της διασφάλισης της επιτυχίας ε, του ΙΤΕΡ σε εύλογο κόστος για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο και με αποδεκτούς κινδύνους η Κομισιόν έχει ε, θεσπίσει ορισμένους, ορισμένους όρους μεταξύ αυτών ε, λογικό, ρεαλιστικό δηλαδή πλαίσιο εκτίμησης του κόστους και ούτε καθεξής. Το Νοέμβριο 2009 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανέλαβε την ομόφωνη υποστήριξή του στο πρόγραμμα ITER με σημαντική αύξηση κόστους εφόσον όμως τηρούνται αυτές οι, ε, αυτοί οι πλαίσια. Ε, συνεχίζει η Επιτροπή ε, να εργάζεται ώστε να διασφαλίζει την τήρηση αυτών των όρων και για το κόστος που έχουν οι σχετικοί όροι εξεταστεί εξαντλητικά με την βοήθεια εθνικών εμπειρογνωμόνων και έχουμε τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις αυτή τη στιγμή που ανέρχονται σε 7,2 δις ευρώ κόστος για την Ευρώπη για την φάση κατασκευής του ίτερ που υπολογίζεται να είναι μέχρι το 2020. γίνονται ε, γίνεται, προωθούνται τα σχέδια αυτά μαζί με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων. Έχει βελτιωθεί τώρα το χρονοδιάγραμμα τον Νοέμβριο του 2009 έγινε νέα εκτίμηση του κόστους και των κινδύνων προς τα κάτω. Φαίνεται πάντως τώρα να είναι τεχνικώς αποδεκτό για την Ευρώπη το σχέδιο. Και σε ό,τι αφορά την ορθή διαχείριση του σχεδίου, ε, ανέλαβε, την Ευρω... ανέλαβε η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή την πρωτοβουλία να κάνει τη σχετική ε, δήλωση και το 2009 με την πρόβλεψη ότι θα χρειαστεί να γίνουν σημαντικές αλλαγές στον οργανισμό του οργανισμού, στο, στον οργανισμό του ΙΤΕΡ Αρχές Ιανουαρίου του 2010 ε, ο νέος διευθυντής κ. Μπρίσκο που βρίσκεται εδώ δίπλα μου διορίστηκε και θα αρχίσει την αναδιάρθρωση του οργανισμού. Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Συμβούλιο του ε, Ιουνίου του 2009 θέσπισε την ε, εκτίμηση για τον οργανισμό που λέει καθαρά ότι οι αλλαγές θα χρειαστούν και στο top management αλλά και στην οργανωτική δομή. Οι απαραίτητες αλλαγές για το top management έχουν ήδη γίνει και για την οργανωτική δομή θα γίνουν τις επόμενες εβδομάδες. Εξέδωσε ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την διαβίβαση και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Στην ανακοίνωση αυτή Το βασικό μήνυμα είναι ότι για να δαπανηθούν με υπεύθυνο τρόπο τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης οφείλουν να διασφαλίσουν ότι το έργο προχωρεί ορθά, με τη σωστή κατεύθυνση και έχει την απαραίτητη χρηματοδότηση για ολόκληρη τη διάρκεια του κατασκευής και λειτουργίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσει ξανά παρόμοια διαδικασία όπως έγινε με τον Γαλιλαίο. Αυτό το λεγόμενο bricolage approach είναι κακό για την βιωσιμότητα του ε, σχεδίου. Και είναι κακό και για τις σχέσεις μας με τους διεθνούς εταίρους μας. Με τους διεθνείς, συγγνώμη, εταίρους μας. Οι χώρες μέλη οφείλουν να αναγνωρίσουν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την ε, διασφάλιση των μακροπρόθεσμων ε, υποχρεώσεων του ΙΤΕΡ και να χορηγήσουν την απαραίτητη χρηματοδότηση για ολόκληρη την φάση ε, κατασκευής και λειτουργίας του. Οι διεθνείς εταίροι μας αναμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει την έγκριση από το Συμβούλιο ΙΤΕΡ της λεγόμενης baseline, που σημαίνει τον στόχο του έργου το χρονοδιάγραμμα και το συνολικό κόστος. Η έγκριση αυτή αναμένεται να γίνει στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου ΙΤΕΡ ε, μέσα Ιουνίου στην Κίνα. Η Κομισιόν θεωρεί ότι μπορεί μόνο να υποστηρίξει την έγκριση της baseline εφόσον έχει λάβει την πολιτική ε, εξασφάλιση από το Συμβούλιο ότι θα υπάρξει μακροπρόθεσμη υποστήριξη ώστε να είναι αξιόπιστη η Ευρωπαϊκή Ένωση ως εταίρος του παγκόσμιου επίπεδο. Η υλοποίηση του ίτερ είναι σημαντική και δεν μπορεί να γίνει ευλόγως σε βάρος των προτεραιοτήτων της Ευρώπης του 2020. Οποιαδήποτε λύση δοθεί θα πρέπει να σέβεται την αρχή αυτή. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του έργου, με 1,4 δις ευρώ στην διάρκεια του 2012 έως 2014. Μιλώ για πιστώσεις υποχρεώσεων. Η Κομισιόν θα είναι έτοιμη να υποβάλει επαρκείς προτάσεις όταν θα έχει ρυθμιστεί το θέμα της μακροπρόθεσμης ανάληψης υποχρεώσεων που θα λάβουν υπόψη όλες τις δυνατότητες χρηματοδοτήσεων σύμφωνα με την διαθεσμική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία και την ορθή δημοσιονομική διαχείριση και σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βεβαίως και ε, με τήρηση των προβλεπωμένων για την Ευρώπη 2020. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ το λόγο κύριο Σπρίσκο για την παρουσίαση του. Καλησπέρα σας κύριε και κύριοι. So I will continue. Sí. Um... Μπορώ να συνεχίσω. Ε, εντάξει. Λοιπόν, Καταρχήν θα ήθελα να διεξηγήσω ότι έχω διαθέσει μια παρουσίαση πριν από τη συνεδρίαση. Μετά μου ζητήθηκε όμως να συγκεντρώσω την προσοχή μου περισσότερο στα θέματα του κόστος και τώρα έχω μια πιο σύντομη παρουσίαση για το θέμα αυτό. Μπορώ όμως να απαντήσω σε ερωτήσεις πάνω στο υλικό που σας έχει αποστολεί. Λοιπόν, πρώτον, δύο λόγια για να σας εξηγήσω τι είναι το ITER. Είναι ένα μηχάνημα για να καταδειχθεί η επιστημονική και τεχνολογική δυνατότητα εφαρμογή ελεγχόμενης σύνδεξης για την παραγωγή ε, ενέργειας. Και βλέπετε εδώ μια εικόνα, είναι μια, ένα τεράστιο μηχάνημα ηλεκτρολογό. Prego. No, I think we, we have, uh, this is... Κοίταξε. Αυτό είναι οργανωμένο για να μπορούμε εμεί να υποβάλουμε ερωτήσει. Ξέρουμε τι είναι το ΙΤΕΡ. Δεν μα ενδιαφέρουν όλα αυτά. Να υποβάλουμε κατευθείαν ερωτήσει. Scusate, sorry. Prego. Prego. C'è una presidenza che risponde. Prego. Eh, consentiamo al nostro ospite di. Ας επιτρέψουμε στον προσκεκλημένο μας ε, να κάνει μια παρουσίαση ε, μπαίνοντας στην ουσία του ζητήματος, γιατί πραγματικά γνωρίζουμε το θέμα. Άρα μπορείτε να επιταχύνετε το ρυθμό σας. Yes. So I won't take... Λοιπόν, δεν θα καταλαβαίνω ιδιαίτερα πολύ χρόνο. Απλώς θα σας δώσω μια εικόνα του Ίντερ και βλέπετε πόσο μεγάλο και πολύπλοκο είναι αυτό το μηχάνημα. Ποιος συμμετέχει στην Ιντερ. Ο συνάδελφος Οκτάβιο Κιντανατριάς εξήγησε ότι πρόκειται για μια διεθνή συνεργασία μεταξύ αυτών των κρατών που αναφέρονται στην εικόνα. Πώς θα κατασκευαστεί το ίτερ είναι σημαντικό για να καταλάβουμε το θέμα του κόστους. Τα διάφορα μέρη του μηχανήματος έχουν κατανεμηθεί σε 85 δέσμες που έχουν κατανεμηθεί μεταξύ των 7 ενδιαφερομένων μερών όπως φαίνεται στη δεξιά μεριά αυτής της εικόνας. Οι περισσότερες συμβολές στο ε, ΙΤΕΡ είναι σε είδος και όχι σε ρευστό χρήμα. Σας δείχνω αυτή την εικόνα του ΙΤΕΡ με ορισμένα από τα βασικά ε, τμήματα που θα πρέπει να δώσει η Ευρώπη μαγνήτες, τμήματα του, του, του δοχείου κενού, τμήμα του πρώτου τείχους και την δομή του κάτω τμήματος του αντιδραστήρα, όπου θα πρέπει να του μεγάλες ποσότητες ε, θερμότητας. Εδώ είναι μία εικόνα καλλιτέχνη, πώς θα φαίνεται το ίτερ μετά από 10 χρόνια δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η εργασία στα οικόπεδα εκείνα. Θα πρέπει να αρχίσει κανονικά τον επόμενο μήνα με την ε, κατασκευή του πρώτου κτηρίου και του υπογείου του μεγαλύτερου κτηρίου αυτή τη στιγμή στην εικόνα. Έχουν ήδη δοθεί οι διάφορες συμφωνίες. Τώρα, για το θέμα του κόστους. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η κατασκευή του ΙΤΕΡ είναι ένα σχέδιο προφανώς τεράστιο μεν και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στους τέσσερις συνήθεις πτυχές ε, του σχεδίου, το εύρος, το χρονοδιαγράμμα, το κόστος και το κίνδυνο. Το γεγονό είναι ότι όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Αν κανένας προς προσπαθήσει να επιταχύνει το χρονοδιάγραμμα, το σημαίνει ότι αυξάνεται το κόστος. Επίσης σας δείχνω εδώ πώς είναι κατανεμμένες οι ευθύνες μεταξύ των διαφόρων υπευθύνων οργανώσεων. Η η οργάνωση ITER στο ΚΑΤΑΡΑΣ, το, η ομάδα δηλαδή, είναι υπεύθυνη για το design και για το εύρος αυτό καθ' δηλαδή το τι χρειάζεται και τι συμπεριλαμβάνεται στο μηχάνημα. Το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή είναι επίσης σε μεγάλο ποσοστό στην ευθύνη της οργάνωσης του ΙΤΕΡ. Εν αντιθέσει προς αυτό, το κόστος και ο κίνδυνος είναι κυρίως στα χέρια του Σύνδεξη για Ενέργεια και άλλων οργανώσεων, ιδίως των οργανώσεων που δίνουν τον εξοπλισμό και συμβάλλουν και σε μετρητά προς το, τη διεθνή ομάδα. Δεν νομίζω ότι οι αριθμοί εκεί μπορούν να... <laughs> ότι είναι πάρα πολύ ορατοί από εκεί που κάθεστε. Είναι ευθυγραμμισμένοι όμως με τα αριθμητικά στοιχεία που υπάρχει στην ανακοίνωση που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινοβούλιο και καταδεικνύουν την εξέλιξη του κόστους από τις εκτιμήσεις του 2001 μέχρι την σήμερα. Και καταδεικνύεται πώς κατανέμεται το κόστος αυτό μεταξύ των συμβολών σε είδος, των συμβολών σε μετρητά και ούτω καθεξής. Μπορούμε αν θέλετε να επανέλθουμε σε οποιαδήποτε λεπτομέρεια θέλετε αργότερα. Τώρα, έχω εδώ μία εικόνα που δείχνει ορισμένους από τους λόγους γιατί αυξήθηκε το κόστος που ανέφερε ο Κταβικιντάνεκτρίας για να δείτε γιατί αυξήθηκε το κόστος για να μπορούμε να το ελέγξουμε από εδώ και πέρα. Κυρίως το design του 2001 δεν ήταν πλήρες. Τα κενά έχουν τώρα ε, πληρωθεί. Και το ξέραμε αυτό γιατί δεν υπήρχε χρόνο. Δεύτερο, το Design του 2001 ήταν πολύ γενικό όσον αφορά την τοποθεσία. Είχε γίνει σε σχέση με οδήποτε τοποθεσία σε όλο τον κόσμο και τώρα χρειάστηκε να προσαρμοστεί για το κάνταρας. Παραδείγματο χάρη εκεί υπάρχουν που και που σεισμοί και γι' αυτό τα κύρια κτίρια θα πρέπει τώρα να κατασκευαστούν σε σεισμικούς ε, μονοτές. Τρίτον, το κλικό δεσάν είχε πάρα πολλούς κινδύνους και γι' αυτό προσθέθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία για να μειωθούν οι κίνδυνοι αυτοί. Αυτό βέβαια οδήγησε σε πληρότερο κόστος. Τέταρτος λόγος, ο πληθωρισμός όσον αφορά τα υλικά από τα οποία κατασκευάζεται το μηχάνημα αυτό, ορισμένα μέταλλα ιδίω, ήταν πολύ υψηλότερη από αυτή που είχαμε κατά νου στις πρώτες εκτιμήσεις κόστους. Σημείο 5. Όπως προανέφερα, το design του 2004 του 2001 συγγνώμη, δεν ήταν ολοκληρωμένο και γι' αυτό έπρεπε να πραγματοποιηθεί περισσότερη εργασία. Χρειάστηκε λοιπόν περισσότερες αμοιβέ εμπειρογνωμών. 6. Πολλές από τι οργανώσει που ασχολούνται με το σχέδιο αυτό είναι τελείως καινούργιες. Ιδίως η οργάνωση του ΙΤΕ στο Κάνταρατς... η Σύνδεξη για Ενέργεια στη Βαρκελόνη και άλλες οργανώσεις σε κάποια άλλα μέρη και χρειάστηκαν τρία χρόνια για να εγκαθιδρυθούν αυτές οι οργανώσεις, να ολοκληρωθούν, να αποκτήσουν το προσωπικό, να γίνουν λειτουργικές. Και γι' αυτό το χρονοδιάγραμμα έχει τώρα μια καθυστέρηση τριών έως τεσσάρων ετών και αυτό επίσης αυξάνει το κόστος. Και τέλος, ο ρυθμός των μερών αυξήθηκε σχετικά με το 2001 και αυτό ε, σημαίνει ότι αυξάνεται το κόστος γιατί υπάρχουν πιο πολύπλοκες διασυνδέσεις μεταξύ τόσων μερών. Τώρα πόσο ισχυρές ήταν οι εκτιμήσεις που υπήρχαν του κόστους. Καταρχήν οι εκτιμήσει κόστου αναθεωρήθηκαν από ανεξάρτητα σώματα πολλές φορές και για το, την ε, οργάνωση ήδη και για την F4E, ε, e συνδεξη για την Ευρώπη. Επίσης, έχουμε να πούμε ότι το κόστος έχει τώρα σταθεροποιηθεί. Οι κύριες αυξήσεις ήδη παρουσιάστηκαν το 2008 και 2009. Από τότε έχουν υπάρξει μόνο πολύ μικρές αυξήσεις για συγκεκριμένους λόγους. Τρίτο σημείο. Έχουμε προχωρήσει τώρα στη συγκεκριμένη φάση αγορών από τη βιομηχανία. Οι αγορέ μέχρι στιγμή είναι λίγο πολύ ευθυγραμμισμένε με τι εκτιμήσει του κόστου. Ορισμένε είναι πιο ψηλέ, ορισμένε κάποιε πιο χαμηλέ, αλλά σε μέσο όρο δεν έχουν διαφορετηθεί, δεν έχουν πολύ. Ε, Επίσης έχει προχωρήσει το σχέδιο, η φάση του design έχει ολοκληρωθεί, υπάρχει μικρότερος κίνδυνος για την ολοκλήρωση. Επίσης είχαν συμπεριληφθεί επιφυλακτικότητες στις εκτιμήσεις για να καλυφθούν πολύ κίνδυνοι στην φάση της παραγωγής και της ε, κατασκευής. Και τέλος δεν υπάρχει πια ανάγκη να υπάρχει ένα περιθώριο για αφύσικους κινδύνους. Τέλος, τελική εικόνα. Ε, αναφέρω ορισμένε ορισμένες δράσεις που ήδη έχουν εισαχθεί για να περιοριστεί το κόστος. Θα πρέπει τώρα να ενδυναμωθούν οι δράσεις αυτές για να μην αυξηθεί περισσότερο το κόστος. Αυτό είναι η τελική εικόνα. Πρώτον, λόγω του μείγματος ευθυνών μεταξύ της οργάνωσης Center και των τοπικών ε, οργανώσεων όπως τη Σύνδεξη για την Ευρώπη θα συνεργαστούμε πιο στενά με την οργάνωση του Ίντερ για να μην αυξηθεί το κόστος ε, με αλλαγέ στα χρονοδιάγραμμα ή στο ευρώ. Δεύτερον, θα αναζητήσουμε δυνατότητε εξοικονομήσει σε όλη μα την εργασία και όπου υπάρχει κάποια αύξηση κόστου, όταν παραδείγματο χρησιμοποιούμε προσφορά για κάποια εργασία ή κάποιο υλικό, θα το αντιμετωπίσουμε έντονα εάν υπάρχει έντονη αύξηση του κόστου. Θέλετε να σταματήσω εδώ και να περάσουμε στις ερωτήσεις. Ωραία, θα σας το αφήνω λοιπόν στην οθόνη αυτό για να το βλέπετε. Σα ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Η πρώτη ερώτηση. Ευχαριστώ Ζητάτε την υποστήριξη όλων των θεσμικών οργάνων, αλλά για να έχετε την υποστήριξή μας θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη. Το 2001 έγινε μία εκτίμηση από εμπειρογνώμονες. Μιλήσατε για 2,7 δις και το 2009 μας ε, μιλάτε για 5,7 δις. αν είχαμε ένα 30% διαφορά, τότε θα το δεχόμασταν. Γιατί εάν υπάρχουν ε, σεισμοί στο Καντεράς, υπάρχουν και στην Ιαπωνία. Μιλάτε για αύξηση του κόστους του προσωπικού ή υποτιμάτε το αρχικό κόστος ή δεν ξέρω τι συμβαίνει. Το ίδιο αφορά το ΠΕΡ της Φιλανδίας. Μας ε, πουλάτε ένα ίτερ, το υποτιμάτε στην αρχή για να γίνει αποδεκτό από την Ευρώπη και στη συνέχεια μας λέτε «Α, υπάρχει μία υπερεκτίμηση». Δεν με τα στοιχεία σας. Όταν δω τα στοιχεία παροπλισμού και λειτουργίας 5 δις, τότε δεν έχουν υπερτιμηθεί. Άρα τα λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα παροπλισμού είναι της τάξης των 5 δις. Γιατί σε λίγα χρόνια θα μας πείτε ότι ε, υπάρχει ένα πολλαπλάσιο κόστος. Θα ήθελα το ελεγκτικό συνέδριο να κάνει μια εκτίμηση του κόστου ΣΥΤΕΡ. Διαφορετικά θα ε, επιβληθούν, θα επιβληθεί το κόστος σε όλα τα κράτη-μέλη. Από αυτή την ε, άσπρη φάλαινα, λέει ο Μιλήτρη, από αυτό το Moby Dick. Köszönöm, Üdvözlöm, tisztelettel üdvözlöm a vezérigazgató urat és az igazgató urat, és köszönöm a... Σας ευχαριστώ, πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε Γενική Διευθυντά. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Εγώ δεν συμφωνώ με τη συνάδελφο που μίλησε πριν από μένα, γιατί νομίζω εδώ συζητάμε για θέματα έρευνα και στην έρευνα θα πρέπει να ε, λαμβάνουμε υπόψη μας κάποιες πτυχές και κάποιους μηχανισμούς. Άμα δούμε πόσα χρήματα χρησιμοποιούσαν πριν από 10 χρόνια για το πρόγραμμα πλαίσιο, θα πρέπει να θεωρήσουμε αυτά τα στοιχεία ρεαλιστικά. Εγώ υποστηρίζω το σχέδιο αυτό. Ζούμε σε περίοδο ενεργειακής κρίσης και για να έρθει η κρίση αυτή χρειαζόμαστε μια ενεργειακή στρατηγική για τους Ευρωπαίους που θα τους βοηθήσει να έχουν ασφαλή τροφοδότηση με ενέργεια. Το σχέδιο ΙΤΕΡ έχει ακριβώς αυτόν τον στόχο και ε, καταδεικνύει ένα παράδειγμα πώς είναι δυνατόν η πυρηνική ενέργεια να χρησιμοποιηθεί και για ειρηνικούς στόχους. Πρόκειται για μια καθαρή πηγή ενέργειας που δεν οδηγεί σε παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα Εκτός από την Κίνα, την Ιδία, την Ιαπωνία και τη ΣΥΠΑ, η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να παίξει ηγετικό ρόλο. Γι' αυτό το σχέδιο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για εν μέρη πολιτικό θέμα. Από όσο ξέρω, αυτό το σχέδιο είναι το μόνο προ... σχέδιο έρευνας που συντονίζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεχθούμε αβέβαιοι την περίπτωση αυτή, τότε ένας από τους εταίρους μας θα μπορεί να μας αντικαταστήσει. Χρειαζόμαστε βέβαια συμπληρωματικές πηγές ε, χρηματοδότησης, αλλά θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες που θεωρούμε καλύτερες. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν μου φαίνεται ότι είναι καλή λύση ούτε η αναδιάρθρωση των δημοσιονομικών πόρων γιατί αυτό θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2020, τη στρατηγική τη γι' αυτό. Εγώ είμαι υπέρ μια λύση που θα δώσει τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη να υποστηρίξουν από κοινού αυτό το σχέδιο. Τα 27 κράτη-μέλη και η Ελβετία θα πρέπει να χορηγήσουν 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ για το σχέδιο αυτό. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της λύσης το σχέδιο ΙΤΕΡ είναι μια πολύ θετική πρωτοβουλία και θα μπορούσε να αποτελέσει καλό παράδειγμα στον τομέα της έρευνας για την ατομική ενέργεια. Πριν από λίγο χρόνο επισκέφθηκα το Ινστιτούτο Κάιτα στην Καστρού και θα ήθελα ο κ. Γενικός Διευθυντής να μας πει πώς είναι το χρόνο. Allora, cogliendo il suggerimento del collega Turco. Χωρίζουμε σε δύο μπλοκ. Οι διερμηνείς θα μείνουν λίγο περισσότερο. Ρεμέκ οντί. Και μετά απαντήσεις και μετά ο άλλος γύρος ερωτήσεων, ο επόμενος γύρος ερωτήσεων. Ja, vielen Dank. Ähm, ich muss sagen... Ευχαριστώ. Κάνω ένα πρώτο σχόλιο πριν να ρωτήσω. Με εκπλήσει που ακούω ότι το 2001 εγκρίθηκε εδώ η πρόθεση ενός σχεδίου του αντιδραστήρα αυτού, μάλλον ε, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ενός σχεδίου του αντιδραστήρα αυτού και μαθαίνω τώρα ότι αποφασίσαμε να χρηματοδοτήσουμε ένα σχέδιο αντιδραστήρα το οποίο δεν ήταν ολοκληρωμένο, δεν ήταν έτοιμο. Εγώ το βρίσκω αυτό σκανδαλώδες. Οι συνάδελφοί μου εδώ που απεφάσισαν τη χρηματοδότηση αυτή, σε ποια βάση αποφάσισαν. Νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη να εξηγήσετε περισσότερο. Αυτό που με ενδιαφέρει πάντως προκειμένου είναι γιατί το Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω δεν μπόρεσε να συνεννοηθεί να συμφωνήσει επί περαιτέρω χρηματοδοτήσεως. Θέλω να μάθω ποια είναι τα σενάρια κόστους που έχει συντάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ποιες πιθανές περιπτώσεις δηλαδή και αν έχει συζητηθεί ένα ενδεχόμενο σενάριο για μια αναβολή εάν δεν έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο, ο σχεδιασμός δηλαδή. Ή εάν πρόκειται να γίνει μια μειωμένη εφαρμογή, μια περιορισμένη εφαρμογή της ε, προσπάθειας αυτής, εάν ενδεχομένως το έργο εγκαταληφθεί, διότι αυτού του είδους η αύξηση του κόστους οφείλει να θέσει και τέτοια ερωτήματα. Ποια σενάρια λοιπόν έχει συντάξει και υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με ενδιαφέρει επίσης και πώς θα συνεχίσει η προσπάθεια αυτή. Θα υπάρξει άλλο Συμβούλιο Ανταγωνισμού το οποίο θα συζητήσει και αν δεν γίνει τέτοιο Συμβούλιο Ανταγωνισμού το οποίο να αποφασίσει για την περαιτέρω χρηματοδότηση τότε θα αναβληθεί το Συμβούλιο Ήτερ ή εν πάση περιπτώσει τι άποψη έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έδωσα το λόγο στο συνάδελφο Ρεμέκ. Έγινε λάθος. Έχετε το λόγο. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ. Εγώ δεν θα κάνω σχόλια, λέει ο κύριος Ρέμεκ. Μία ερώτηση μόνο. Ένα σύντομο σχόλιο, αν θέλετε. Εγώ θεωρώ ότι το ίτερ αξίζει τον κόπο. Όταν οι άνθρωποι για πρώτη φορά άναψαν φωτιά, φοβήθηκαν. Κιόλας. Φοβήθηκαν μεν, ωστόσο η φωτιά ήταν ένα σημαντικό βήμα για την ανθρωπότητα προς τα εμπρός. Το ίδιο και τώρα. Πιστεύω ότι θα είναι ένα τεράστιο βήμα. Βέβαια, το κόστος έχει αυξηθεί τρομερά. Δεν πρόκειται όμως μοναχά για έργο ευρωπαϊκό. Ποιο είναι ο καταμερισμό τη αύξηση του κόστου και στου άλλου εταίρου οι οποίοι συμμετέχουν στην προσπάθεια. Και ποια είναι η θέση των άλλων εταίρων. Έχουμε δύο παρεμβάσεις ακόμα. Μπριτζίνα e OD. Diamo la parola per una breve replica e poi ancora rapidamente. Μπορείς να απαντήσεις και μετά θα έχουμε το δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Σύντομα να απαντήσετε, αλλά με σαφήνεια. Chi comincia? Prego. Ποιος θα αρχίσει? Mr. Brisco. Risposte brevi, però molto puntuali alle domande che sono state puntuali. Εν συντομία σας παρακαλώ. So perhaps I can uh, start with a question. Μπορώ ίσως να αρχίσω απαντώντας την ερώτηση που τέθηκε σχετικά με τον σχεδιασμό του μηχανήματος. Το 2001 το design ήταν καλό. Ήταν πλήρες το μηχάνημα. Όταν είπα ότι δεν ήταν ολοκληρωμένο, δεν εννοώ ότι ήταν μισοφτιαγμένο. Υπήρχαν κάποια κενά. Όλα τα συστήματα από τα οποία συναπαρτίζεται το μηχάνημα αυτό είχαν σχεδιαστεί, αλλά ιδίως σχετικά με τα interface μεταξύ των συστημάτων και ορισμένες από τις συνδέσεις μεταξύ των συστημάτων δεν υπήρχαν όλες οι λεπτομέρειες. Δεν είχαν σχεδιαστεί όλες οι λεπτομέρειες. Με αυτή την έννοια ήταν ατελές το σχέδιο. Είπα επίσης ότι δεν είχε επιλεγεί η τοποθεσία και το σχέδιο δεν είχε προσαρμοστεί σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Υπήρχε λοιπόν ακόμα, έμεινε ακόμα λοιπόν κάποια δουλειά να γίνει ε, για το λόγο αυτό. Και τρίτο, Το σχέδιο ήταν καλό το 2001, αλλά υπήρχαν ορισμένες πτυχές του που θεωρήθηκε ότι έθεταν σε κίνδυνο ενδεχομένως την τελική λειτουργία του μηχανήματος. Αυτά αναθεωρήθηκαν και έχει τώρα ληφθεί απόφαση να προσθεθούν και άλλα χαρακτηριστικά στο μηχάνημα, ναι, στο, στο μηχάνημα, ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι αυτοί. Τώρα, κατά κάποιο τρόπο, έχει τελειώσει, το, έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο και έχει βελτιωθεί, αλλά οι δράσεις αυτές συνεπάγονται κάποιο κόστος. Αυτό μπορώ να πω για την ώρα. Yes, I Ως προς το σενάριο αυτό, η Επιτροπή ήταν απόλυτα σαφή στην ανακοίνωση. Θέλει μία δέσμευση χρηματοδότηση μέχρι το τέλος της κατασκευής και της λειτουργίας του μηχανήματος. να διασφαλιστεί δηλαδή αυτή η χρηματοδότηση για να μην αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση κρίσης όπως αντιμετωπίζουμε σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι επειδή η εκτίμηση κόστου είναι 7,2 δις, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε αυτή τη χρηματοδότηση μέχρι το 2020 τουλάχιστον για την κατασκευή. Για τη λειτουργία δεν υπάρχει λόγος για αύξηση του κόστους. Η κατασκευή χρειάζεται νέα υλικά, αλλά ε, μιλάμε και για την συντήρηση και για το προσωπικό που θα ασχοληθεί με αυτήν, καθώς και τον παροπλισμό της μηχανής, του μηχανήματος. Άρα δεν έγινε μία επανεκτίμηση εδώ, γιατί θεωρούμε ότι όλα αυτά εντάσσονται στο σενάριο που έχουμε προβάλει. Άρα μέχρι το 2020 έχουμε μία δέσμευση και εάν την αναλάβει το Συμβούλιο, η Επιτροπή θα παρουσιάσει μία πρόταση για τις ενδεχόμενες επιλογές για την χρηματοδότηση το 2012-2013 που υπάρχει αυτό το χάσμα μεταξύ του προϋπολογισμού μας και του επιπρόσθετου κόστους που επιβάλλεται. Ως προς το χρονοδιάγραμμα, έτσι έχει το χρονοδιάγραμμα, τώρα είμαστε στη φάση κατασκευής η οποία άρχισε. Τώρα αρχίζουν οι διαγωνισμοί για τις κτηριακές εγκαταστάσεις τους επόμενους μήνες. Θα γίνει ε, καταμερισμός σε 12 διαγωνισμούς. Θα γίνει η συγκρότηση το 2015. Και το τέλος της κατασκευής, το πρώτο πλάσμα, όπως λέγεται, θα είναι έτοιμο το 2019 αρχή του 2020 και το 2026-2027 θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα των αντιδράσεων. Εντάχει, ο Merci, Madame la Présidente. Je voudrais... Euh, Λυπάμαι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία στην ε, απαρχή αυτού του θέματος. Είπατε κύριε Καντάνα ότι τα κράτη-μέλη ήταν συνυπεύθυνα. Όχι, η Κομισιόν ήταν υπεύθυνη. Γιατί το Συμβούλιο σας ε, υπέβαλε ένα ερώτημα, εσείς δεν απαντήσατε και το Μάιο του 2010 μας δίνετε μία σύντομη απάντηση. Δεν υπάρχουν επεξηγήσεις και ευχαριστώ τον Διευθυντή Μπάσκο που έδωσε απαντήσεις. Χωρίς επεξηγήσεις, βλέπετε τι συμβαίνει σε αυτή την Επιτροπή. Έχουμε δημοσιονομικούς περιορισμούς ως προς επιστημονικά ζητήματα ενεργειακά και ούτω καθεξής είναι λυπηρό. Αλλά δίνουμε την εντύπωση ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη και όχι τα κράτη-μέλη. Το λέω γιατί ως προς την κρίση του ευρώ εμείς αμφισβητήσαμε τα κράτη-μέλη γιατί δεν τήρησαν το σύμφωνο σταθερότητας, τώρα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν υπάρχει καμία παράγραφος για την παγκόσμια διάσταση αυτού του project. Δεν είναι ευρωπαϊκό. Είναι παγκόσμια εμβέλειας. Στις δημοσιονομικές δυσκολίες ε, έχετε έρθει σε επαφή με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Ποια είναι η θέση των Αμερικανών στη Σανγκάη, την προηγούμενη εβδομάδα στην Παγκόσμια Έκθεση. Υπάρχει ένα τέτοιο μήνυμα το οποίο κινήσατε και προς τα εκεί. Ποια νομίζει ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που διαχειρίζεται παγκόσμια ζητήματα. Λυπάμαι για την εξέλιξη. Θα ήθελα να το ξαναδεί η Επιτροπή πριν στους συντονιστές. Είπα να έχουμε μια κοινοβουλευτική πρωτοβουλία. Δεν ξέρουμε τι θα αποφασίσουμε. Θα αναλυφθεί μια πρωτοβουλία αλλά πρέπει να ανταποκριθούμε, διότι το 2050 θα έχουμε μία ανθρωπότητα. Εσείς θα ζείτε γιατί είσαστε γυναίκα. Έχω ένα γιο 7 μηνών σήμερα. Θα ζει το 2050, γι' αυτό εργαζόμενοι στις επόμενες γενιές. Grazie. La parola al collega Turmes, poi Brid... Turmes. che deve porre una domanda a lei, dottor Quintana. Um, I have... Τέσσερις συγκεκριμένες ερωτήσεις και αναμένω συγκεκριμένες απαντήσεις. Πρώτη, ποια είναι η συνεισφορά της Γαλλίας, η οποία υποσχέθηκε ότι θα καταβάλει το 20% του κόστους της κατασκευής. Όπως αυτά υπολογίστηκαν τον Μάρτιο του 2010, το κόστος αυτό δηλαδή, αυτά θα πληρώσει, τα 20% από αυτά θα πληρώσει η Γαλλία. Δεύτερη ερώτηση. Μπορείτε να μας προσφέρετε μια ανάλυση ανά χώρα μέλος να δούμε ποιος θα πληρώσει τι, ποιο ποσοστό του πρόσθετου κόστους. Το Λουξεμβούργο για παράδειγμα, η χώρα μου, το Βέλγιο, η Γαλλία, τι θα πληρώσουν όλοι αυτοί, δεν ξέρουμε στους υπολογισμούς σας κάθε μια από τις χώρες μέλη τι θα κληθεί να πληρώσει. Τρίτο, η διεθνής διάσταση. Η κυβέρνηση Ομπάμα στον προπολογισμό του 2011, στον αμερικανικό προπολογισμό του 2011, προβλέπει 80 εκατομμύρια δολάρια για το ίτερ. Δεν είναι διόλου όμως αυτό που θα πρέπει να πληρώσουν σύμφωνα με τους δικούς μας υπολογισμούς τουλάχιστον με αυτές τις προφορίες που έχουμε σήμερα διαθέσιμες επισήμως, ανάμεσα δηλαδή σε αυτά που προβλέπουν οι Αμερικανοί στον προπολογισμό τους και που θα έπρεπε να προβλέπουν, που θα έπρεπε να προβλέπουν κανονικά, λόγω του, της μεγάλης αξίωσης του κόστους. Εν τέλει, πώς τολμάτε, πώς τολμάτε παραλαμβάνω, να αναλάβετε δέσμευση μέχρι το 2020 για όλο το κόστος της κατασκευής δηλαδή. Και εμείς ως Κοινοβούλιο δεν έχουμε ακόμα αποφασίσει δεν έχουμε ακόμα εγκρίνει τη δημοσιονομική προοπτική μετά το 2013. Άρα αυτό που κάνετε στην ουσία, μάλλον ρωτώ, προσπαθείτε να προκαταλάβετε την δαπάνη πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στην, ε, ε, που θα προσκύψουν από την επόμενη συναπόφαση για την δημοσιονομική προοπτική 2013. Ζεντίνα. Ε, υποστηρίζουμε το έργο. Διότι οι ελπίδες που συνδέονται με την πυρηνική σύνδεξη πρέπει να επαληθευτούν. Είναι σημαντικός δρόμος για το μέλλον και θα τονίσω στους προσκεκλημένους μας ότι αυτοί που τους επιτίθεται κυρίως είναι οι πράσινοι οι οποίοι βλέπουν ως κίνδυνο, διότι αν επιτύχει η πυρηνική σύνδεξη, χάνουν το ιδεολογικό τους υπόβαθρο. Εγώ λοιπόν δεν συμφωνώ με την ευρικότητα αυτών των πρασίνων. Σα θέτω ερωτήσει που μπορείτε να απαντήσετε. Εσεί βρίσκεστε μέσα, στα, μέσα στη μέση του σχεδίου. Βρίσκεται στη μέση του σχεδίου. Είναι ε, λοιπόν δυνατόν να απαντήσετε ήδη στι ερωτήσει αυτέ. Αυτό η ερώτησή μου είναι εξή. συνεργάζεστε με το Ρώσο-Ιταλικό σχέδιο που νομίζω ότι λέγεται Ignita. Και τι νομίζετε, αν μπορεί δηλαδή η σύνδεξη να προκύψει μέσα από μια αντίδραση σε ένα λέιζερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ ε, που παραμένετε λίγο ακόμα. Ε, αν δεν μπορέσουν να θα συνεχίσουμε χωρίς διερμηνία. Ο κύριος Ρέμεκ, ποιο είναι το ποσοστό του αυξημένου κόστους που θα αναλάβουν οι άλλοι και θα αναλάβουν κάποιο, διότι βέβαια τότε είναι διαφορετική η εικόνα σε σχέση με το ποσοστό που θα κληθεί να συνεισφέρει η ευρωπαϊκή πλευρά. A tutti, sì, sì, sì. In inglese ormai parliamo solo. Sì, sì, va bene. I'll, I'll speak in English. Let me first address the international issue because... Ως προς το διεθνές ζήτημα, το θίξατε οι περισσότεροι αν όχι όλοι. Αυτό που θα πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι η συμφωνία προβλέπει ότι όλοι οι διεθνείς ε, εταίροι θα συμμετάσχουν στα πλαίσια αυτά. Θα συνεισφέρουν όσο μπορούν. Δηλαδή θα συνεισφέρουν με ένα μέρος τη, τη, της ανάλογα με το συνολικό κόστος. Αν υπάρχει λοιπόν αύξηση του κόστους για την ευρωπαϊκή συνιστόσα δεν είναι πρόβλημα για τους άλλους. Όλοι θα ε, συμμετάσχουν. Κρίναμε αυτά τα συστατικά το 2001. Είπαμε ότι είναι μάλλον ισομερίζουμε το κόστος, συνεισφέρουμε με 45% και οι άλλοι 9% καθένας. Και η Ευρώπη με 45,46% του συνολικού κόστους του μηχανήματος. Αυτό εκτιμήθηκε στην αρχή. Αν έχει τώρα αυξηθεί για κάθε συστατικό διαφορετικά, αυτό αφορά τον κάθε συνεισφορέα. Άρα αν τώρα στην Ευρώπη έχουμε πρόβλημα, είναι δικό μας το πρόβλημα. Οι άλλοι θα έχουν ε, πρόβλημα ως προς τη, τη δική τους συνιστόσα, τη δική τους συνεισφορά. Με τα κτίρια είχαμε κόστος 550 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα στοιχίζουν ένα πολλαπλάσιο, 1,4 δις, 1,3-1,4 δισεκατομμύρια και αυτό το αναγνωρίζουν και οι εμπειρογνώμονες που έρχονται από τα κράτη-μέλη. Οι άλλοι δεν θέλουν να συμπεριληφθούν στην αύξηση αυτού του κόστους. όλοι ανέλαβαν την αύξηση του κόστου στον προϋπολογισμό τους, αλλά το επίπεδο ε, συνεισφοράς είναι πολύ υψηλότερο από ό,τι τώρα. Και η δική μας ε, εισφορά βρίσκεται στην αρχή. Συνεισφορά. Και όπως καταλαβαίνετε το κτίριο, οι κτηριακές εγκαταστάσεις είναι το πρώτο που μας απασχολεί και είναι υπό τη δική μας ευθύνη. Οι διεθνείς εταίροι αντιμετώπισαν αύξηση κόστους, αλλά όχι όπως εμείς. Όλοι οι άλλοι εταίροι θα ήθελαν και εμείς να υπογράψουμε, να εγκρίνουμε αυτή την κατευθυντήρια γραμμή, αλλά δεν θα το κάνουμε εάν δεν υπάρχει δέσμευση χρηματοδότησης. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αν δεν έχουμε την χρηματική υποστήριξη. Κύριε Τούρμες, ως προς τη συνεισφορά των ΙΠΑ, διακόπτει η Πρόεδρος. Κάτι ελέγχθη εκτός μικροφώνου. Ως προς τη διεθνή διάσταση, η συνεισφορά των ΙΠΑ ως προς συμφορά των έχουν εγγράψει 2,2 δις δολάρια για ολόκληρη την κατασκευή. Είναι το δικό τους μερίδιο. Δεν ξέρω πώς το υπολόγισαν. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά τα στοιχεία. Um, and it's true that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 αυτό ευχαριστώ. πολύ